Okay, Ας ξεκινήσουμε. Καλημέρα. Να αφήσουμε τον κύριο Λάιφρυ να ξεγλιστρήσει απαρατήρητος από την πόρτα. Κύριος Λάιτφριντ. Ας ξεκινήσουμε με ανακοινώσεις του Προέδρου και να καθορίσουμε συντάκτες και συγγητές. Αυτά που συζητήσαμε στους συντονιστές χτες. Όσον αφορά το διορισμό εισηγητών, έχουμε συμφωνήσει όσον αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύμβαση για τις διεθνείς μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων που τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του Βίλνιους Αυτή ήταν η συμφωνία του Μαΐου του 1980. Μάλλον θα την αναλάβει ο Πρόεδρος. Αυτό αποφασίσαμε οι συντονίστες. Το ίδιο όσον αφορά ε, τη μεταφορά εξοπλισμού, μεταφορά εμπορευμάτων υποπίεσης. Υποπίεση. Μετά έχουμε ανακοινώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έκθεση προόδου για την εφαρμογή τη οδηγία ασφάλεια των σιδηροδρόμων και την οδηγία για τη διαλειτουργικότητα. Ελπίζω να συμφωνείτε κι εσεί. Είπαν οι συντονιστέ να υποβληθεί προφορική ερώτηση με συζήτηση. Να υποβληθεί ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέταρτο, ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ολοκληρωμένη πολιτική για θαλάσσιες μεταφορές για καλύτερη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο δεν εμπεριέχει πολλά στοιχεία μεταφορών και ελάχιστα θαλασσίων μεταφορών παρά τον τίτλο. Λίγα πράγματα θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Για τις γνωμοδότησεις έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις. Η πρώτη αφορά την απαλλαγή του 2008, του Γενικού Προπολογισμού του 2008, κεφάλαιο 3, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σύμφωνα με το κανονικό μας σύστημα κυκλικής αναλλαγής, η ομάδα S&D ε, θα καθορίσει συντάκτη, ωράριο εργαζομένων στις οδικές μεταφορές, ψήφισε στις 29 Σεπτεμβρίου Επιτροπή Μετα... να μην απορρίψει την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά να συντάξει νέα έκθεση. Η κυρία Μπάουερ του ΕΛΚ είναι η νέα εισηγήτρια. Εγώ προτείνω ότι εφόσον η Επιτροπή Απασχόλησης θα ετοιμάσει νέα έκθεση, εγώ θα έλεγα να ετοιμάσουμε μια γνωμοδότηση επί του θέματος. Οι συντονιστές συνεφώνησαν και βάσει του συστήματος εκπεριτροπής αναλήψεως η ομάδα S&D είναι εκείνη που θα αναλάβει το θέμα. Είσαστε όλοι ευτυχείς με αυτά. Μάλιστα. Καλώς. Σχέδιο δράσης για αστική κινητικότητα. Στις 30 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε σχέδιο δράσεως για την αστική κινητικότητα και εν τη απουσία της καθυστερημένη εκθέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να σα πω ότι το Κοινοβούλιο υιοθέτησε έξι ιδέε πρωτοβουλία τον Απρίλιο ενεστώτος έτου. Ο Ζιλ Σαβαρή ήταν ο εισηγητής. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουμε εργασίες επί άλλης εκθέσεως ιδίας πρωτοβουλίας εντός 12 μήνου. Άρα επιτρέπεται να ξεκινήσουμε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας επί του δύο θέματος τον Απρίλιο του 2010. Γι' αυτό έχουμε κάποιο δίλημα. Οι συντονιστές σας συστήνουν να διεξαχθεί συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανείς δεν μας εμποδίζει να το κάνουμε αυτό. Να το συζητήσουμε το θέμα και διαδικαστικά να αξιολογήσουμε τη δυνατότητα μια, ενός ψηφίσματος που θα συνοδεύει αυτή την προσπάθεια. Απαγορεύει ο τουρκικός κανονισμός νέα έκθεση μέχρι τον Απρίλιο του χρόνου, αλλά ο εξωτερικός κανονισμός δεν απαγορεύει συζήτηση και ενδεχομένως ένα συνοδευτικό ψήφισμα. Η σύσταση των συντονιστών είναι αυτό να κάνουμε. Σας ικανοποιεί? Τέλεια! Ακροάσεις και αντιπροσωπείες. Οι συντονιστές προτείνουν τις κάτωθοι αντιπροσωπείες. Τέσσερις αντιπροσωπείες. Σλοβενία, Κροατία, Αυστρία. Ανταλλαγή πρακτικών όσον αφορά α, τις μεταφορές με διάφορους τρόπους μεταφορών σε αυτές τις χώρες. Ανταλουσία, ομάδα S&D. Λετωνία, Εστονία, ανάπτυξη του Βαλτικού Σιδηροδρόμου και σημείων διέλευση στα σύνορα με τη Ρωσία. Η ECR και η ALDE ήθελαν το θέμα και συμφώνησαν να συνεργαστούν και από τους πρασίνους νοτιοανατολική τσεχική α, α, Τσεχία, Σλοβακία και άλλες υποδομές και διασυνδέσεις και βλέπετε ότι εδώ έχει αναμειχθεί ο Μάικλ σε όλα αυτά και αφορά τον βιώσιμο τουρισμό αυτή η ομάδα τον αναλαμβάνει. Επίσης υπάρχει μια δυνατότητα συνάδελφοι να συγχωνευθούν οι προσπάθειες του ΕΛΚ και των Πρασίνων. Ζήτησα από τις δύο ομάδες να προσπαθήσουν να συνεννοηθούν αν μπορούν να συγχωνεύσουν τις εργασίες τους. Άρα θα έχουμε τρεις μεγαλύτερε αντιπροσωπείε αντί τέσσερι μικρότερε. Αν δεν το κάνουν αυτό θα έχουμε τέσσερι μικρότερε αντιπροσωπείε. Λοιπόν, θεωρήστε ότι έχουμε τέσσερι μικρότερε αντιπροσωπείε, αρέσει τελικά να έχουμε τρει μεγαλύτερε αντιπροσωπείε που θα είναι καλύτερο αυτό. Επίση υπάρχει και αντιπροσωπεία ψηλού επίπεδου που θα επισταθεί τέσσερα κάτι μέλη. Μάλλον θα πάνε τετραμερεί, θα πάνε στη Ουάσιγκτον αρχέ του επομένου έτου για να αναμειχθούν στη φάση των υπραγματεύσεων στου ανοιχτού ουρανού. Υπάρχουν τίποτα παρατηρήσεις. Όχι. Όσον αφορά τις ε, ακροάσεις, ζήτησαν οι συντονιστές να ετοιμάσουμε τρεις ακροάσεις. Θα θυμόσαστε τι είπαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση, όπου εκεί τι είχαμε πει. Αντί να έχουμε τέσσερις μεγάλες ακροάσεις, να έχουμε συνεδριάσεις μελετών και να ακούμε πυρογνώμοντες, αντί να έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ε, μέλη των ε, ομάδων πίεσης ε, των διαφόρων τομέων να παρίστανται. Θεώρησαν όμως ότι χρειαζόμαστε τρεις ακροάσεις. Έχουμε μία ακρόαση για τη οδική ασφάλεια που συνδέεται με το σχετικό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το εξωτερικό κόστος για τα πλοία και παροχή ενέργεια στα λιμάνια, συμβολή στην καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο. Ο κύριο Ντερόιτε μπορεί ενδιαφέρεται και ε, αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας, προκλήσεις στο μέλλον και προπτικές που έχουν τα νησιά και απομονωμένες περιοχές. Άρα έχουμε ε, δύο θαλάσσια ε, θέματα και οδικές ασφάλειες ακροάσεις. Για τα άλλα θα πάρουμε ε, αποφάσεις ανάλογα με τις συνεδριά, της, συνεδριάσεις μελέτης. Αυτές είναι οι ακροάσεις λοιπόν. Είσαστε όλοι ικανοποιημένοι. Ωραία υπέροχη αυτή η Επιτροπή τέλο πάντων. Το επόμενο θέμα είναι η Επιτροπολογία. Θα θυμόσαστε ότι πήραμε μία απόφαση να έχουμε δύο μέλη α, για τις Επιτροπές ακολουθώντας τη διαδικασία της Επιτροπολογίας. Βέβαια, προσπα... να μην προσπαθήσω να ξεγελάσουν χρησιμοποιώντα την Επιτροπολογία. Αυτό είναι η προϋπόθεση. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς κατά το παρελθόν και ο κύριος Κουν και ο κύριος Αλκαντράη προτάθηκαν από τους συντονιστές σαν η ε, τσάρη της επιτροπολογίας, η αρμόδια για την επιτροπολογία. Και θα ξεκινήσουμε ε, από τον Νοέμβριο. Ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που έχουν ε, υιοθετηθεί σε πρώτη ανάγνωση, ενημέρωσε τους συντονιστές γιατί αναμένουμε κάποιες κοινέ θέσει του Συμβουλίου. Καμία απάντηση δεν δόθηκε από τον Σουηδό Υπουργό, τη Σουηδό Υπουργό για ένα γράμμα που έστειλα για την Ευρωβινιέτα. Δεν νομίζω θα έρθει κάτι γρήγορα σαν αυτά τα δικαιώματα των επιβατών και θαλάσσιες μεταφορέ και για λεωφορεία και πούλμαν. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή μάλλον στη συνεδρίασή της του Νοεμβρίου, στην Επιτροπή Μεταφορών, για να συζητήσουμε αυτά που θα υποθούν στο Συμβούλιο Μεταφορών τον Οκτώβριο. Και όσον αφορά τα πούλμαν και το λεωφορείο, πιθανότατα το Συμβούλιο να αποφασίσει το Δεκέμβριο. Και όσον αφορά το ITS και το θέμα των διαδρόμων μεταφορών εμπορευμάτων, η Επιτροπή έδωσε εντολή στους εισηγητές να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη Σουηδική Προεδρία. Καλώς! Είσαστε όλοι ικανοποιημένοι. Αν ναι, αυτές είναι οι ανακοινώσεις που είχα. Ποιος είστε? Ο κύριος Βαντάλεν. Ο, ο, Ζήλερ δεν είναι εδώ. Πρέπει... Την επόμενη εβδομάδα παίρνω καινούρια γυαλιά, ξέρετε. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε συζητήσουμε και την επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόβλημα των πιλότων. Κύριε Βαντάλε, δίκιο έχετε. Ε, είπαμε να στείλουμε γράμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας διευκρινήσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογή και τη μελέτη που έγινε όσον αφορά τις ώρες πτήσεων. Αν υπήρχαν επιστημονικές μελέτες ή όχι πάνω στο θέμα. Και συμφωνήσαμε ότι θα κάνω αυτό και θα ε, επανέλθω να ενημερώσω τους ε, συντονιστές όταν θα λάβω κάποια απάντηση. Καλώς. Ωραία. Μετά, επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων με την ΕΜΣΑ, με τον διευθυντή της ΕΜΣΑ, τον κύριο Ντερόιτερ, ο οποίος είναι μαζί μας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Ναυσιπλοείας. Τον ξέρω από παλιά τον κύριο Ντερόιτερ, Ιδιαίτερη χαρά για μένα που είναι εδώ ο κύριος Ντερόιτερ και ήρθε να μας μιλήσει για το έργο της Επιτροπής αυτής Ασφάλισης Αφρικορίας, της ΕΜΣΑ και έχετε το λόγο κύριε Ντερόιτερ. Ευχαριστώ πρόεδρε και καλημέρα σας. κλήθηκα να κάνω μία 15 λεπτή maximum εισαγωγή, το οποίο και θα κάνω, και θα σας δείχνω και κάποιες φωτογραφίες. Δεν είναι ένα, μια παρουσίαση PowerPoint, απλά μια παρουσίαση φωτογραφικά αυτών των συνοπτικών ε, σημείων που σας λέω. Σας ευχαριστώ καταρχάς που μου δώσετε την ευκαιρία να παρουσιάσω το έργο της ΕΜΣΑ σήμερα. Είχαν γίνει πρόσφατα παρόμοιες εμπειρίες και με τους συναδόλφους από τις ε, υπηρεσίες ε, σιδηροδρόμων και αεροπορικών μεταφορών. Και χαίρο που βλέπω ότι η Επιτροπή ενδιαφέρεται τόσο για τις, ε, τους τρεις οργανισμούς μεταφορών. Αξίζει κάτι τέτοιο, διότι όλες, όλοι αυτοί οι οργανισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των κανόνων που εσείς ψηφίζετε εδώ. Βεβαίως, υπάρχει πάντα δυνατότητα καλύτερης και, μεγαλύτερη, και ε, καλύτερης ε, υλοποίησης και μεγαλύτερης βελτίωσης των υλοποιηθήσεων των, των προτάσεων. Η ΕΜΣΑ δημιουργήθηκε στο ξεκίνημα της τωρινής δεκαετίας ως ένα, ένας από τους οργανισμούς ασφάλειας ασχολείται με την υλοποίηση ενός τεράστιου όγκου ε, τεχνικού χαρακτήρα κυρίως νομοθετικών κειμένων, των εργόμενων πακέτο έδικα και ως κανονιστικός οργανισμός έχει ε, μία εντολή σαφώς καθορισμένη που περιλαμβάνεται στους κανονισμούς του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, έχει νομική προσωπικότητα, έχει προπολογισμό δικό της και λογοδοτεί για τις δράσεις ή τις παραλήψεις της. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η γενική πολιτική στον τομέα δραστηριοτήτων μας ορίζεται από την Επιτροπή με την οποία έχουμε μια προνομιούχα σχέση στην οποία θα επανέλθω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εμπλέκεται μεν στην καθημερινή δραστηριότητα του ΕΜΣΑ, αλλά παίζει βεβαίω σημαντικό ρόλο σε όλα τα θέματα που αφορούν τον προπολογισμό και την νέα νομοθεσία το Κοινοβούλιο, ιδίω η Επιτροπή σα, μα βοήθησε πολύ τα τελευταία χρόνια. Ποιε είναι οι βασικέ ευθύνε μα. Καταρχά, το έργο τη ΕΜΣΑ περιλαμβάνεται σε τρει ομάδε, αν θέλετε. Πρώτον, να επικουρεί την Επιτροπή σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του κεκτημένου ασφάλειας για τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και την επικουρία στην προετοιμασία νέας νομοθεσίας. Στο ίδιο πλαίσιο συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές για μια σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή των συχνά σύνθετων κειμένων ε, νομοθετικού χαρακτήρα. Δεύτερο καθήκον, δεύτερη ομάδα καθηκόντων, η ΕΜΣΑ μετά την το ναυάγιο του του πλοίου Πρεστής το 2002, ανέλαβε και επιχειρησιακά καθήκοντα στη θάλασσα, που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρήπανσης. Σήμερα η ΕΜΣΑ έχει 16 σκάφη καθαρισμού ρήπανσης που βρίσκονται σε διάφορα σημεία σε όλη την ακτογραμμή της Ένωσης. Τα κράτη-μέλη μπορούν να καλέσουν τα σκάφη αυτά σε περίπτωση που υπάρχει μείζον απειλή ρήπανσης από πετρέλαιο των ακτών τους. Έχουμε ένα σύστημα διάγνωσης της ε, μέσω δορυφόρου που λέγεται Clean CNET. Τρίτον, η ΕΜΣΑ ανέλαβε την ευθύνη να αναπτύξει και να χειρίζεται κάθε σύστημα πληροφόρησης ε, με στόχο την επίτευξη των στόχων υλοποίησης της οδηγίας παρακολούθησης της κυκλοφορίας. Αυτό που θα πω σε λίγο. Να σας περιγράψω τώρα με λίγα παραδείγματα και με λίγες εικόνες τι σημαίνει, τι σημαίνουν αυτά, τα, αυτές οι τρεις ομάδες καθηκόντων συγκεκριμένα. Πρώτον, επικουρία στην Επιτροπή για την εφαρμογή κτλ. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΜΣΑ διεξάγει πολλές επιθεωρήσεις. Η, επιθεωρή, η προσέγγιση της επιθεώρησης βασίζεται πάντα στην αρχή της, παρα, της επιθεώρησης των επιθεωρητών και του ελέγχου των ελεκτών. Για παράδειγμα, επιθεωρούμε το έργο των εταιριών νεογνωμόνων και αυτή είναι αυτοί που εξετάζουν κατά πόσον η κατασκευή και επισκευή σκαφών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ανώτατα δυνατά με τις ανώτατες δυνατές προδιαγραφές. Επιθεωρούμε αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς Euro Veritas, American Bureau of Shipping, Bureau Register, τους ελεγκτικούς, τις εταιρείες οροκοτών ελεγκτών εντός και εκτός Ευρώπης. Επισκεπτόμαστε ναυπηγεία στην Κίνα και αλλού για να επιθεωρήσουμε, για να εξετάσουμε κατά πόσον οι επιθεωρητές αυτοί κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεύτερο παράδειγμα. Όπως γνωρίζετε, τα περισσότερα θαλάσσια ατυχήματα δεν προκαλούνται από τεχνικό πρόβλημα αλλά από ανθρώπινο λάθος. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΜΣΑ ελέγχει την ποιότητα της ναυτικής κατάρτισης και στα κράτη-μέλη και στις τρίτες χώρες. Τρίτες χώρες, γιατί όπως γνωρίζετε, η πλειοψηφία των ναυτικών που βρίσκονται σε ευρωπαϊκά σκάφη δεν προέρχονται από την Ένωση. Οι ναυτικοί προέρχονται από Φιλιππίνες, από την Ινδονησία, από την Ουκρανία κλπ. Άρα, συνολικά, έχουμε ναυτικούς σε πλοία της Ένωσης από 50 διαφορετικές χώρες εκτός Ένωσης που δουλεύουν στα σκάφη αυτά. Η ποιότητα της κατάρτισής τους πρέπει κατά την άποψή μας να ελέγχεται. Όπως και τα πιστοποιητικά και διπλώματα που λαμβάνουν. Επίσης, ε, σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς ε, Ναυτιλιακού Οργανισμού, το, ε, ο, το κράτος που, ελέγχει, που δέχεται ένα σκάφο, έχει το δικαίωμα να ελέγξει την ποιότητα της κατάρτισης των ναυτικών. Αλλά αν και τα 27 κράτη άρχισαν να πηγαίνουν στις Φιλιππίνες και να ελέγχουν την ποιότητα της εκπαίδευσης των ναυτικών εκεί, θα κόστισε κάτι τέτοιο πολύ. Για λόγους αποτελεσματικότητας λοιπόν αποφασίσαμε ότι η ΕΜΣΑ θα διεξάγει τις δραστηριότητες επιθεωρήσεις εξ ονόματος όλων των κρατών της Ένωσης. Θα μπορούσα να σας πω και περισσότερα πράγματα για την επιθεώρηση, δεν το κάνω. Απλά θέλω να υπογραμμίσω ότι το έργο της επιθεώρησης συνολικά περιλαμβάνει κατάρτιση εκθέσεων που αποστέλλονται στην ε, Επιτροπή η οποία αποφασίζει για τη συνέχεια που θα, που θα ε, δώσει στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο έλεγχο. Βεβαίω, αντίγραφο του, της έκθεσης παίρνει και ο οργανισμός ή το κράτος που δέχεται τον, ε, την ίδια, λαμβάνει επίση την ίδια έκθεση για να προχωρήσει σε βιοθωτικές κινήσεις αν θέλει. Κάποια άλλα παραδείγματα του τι κάνουμε για την Επιτροπή είναι τα εξή. ζητά η Επιτροπή να να, να, να ετοιμάζουμε μελέτες γιατί αυτέ τι μέρε ετοιμάζουμε ένα κείμενο για τι εκπομπέ αερίων του διοξιδίου του άνθρακα από τα σκάφη. Αλλά κάνουμε και μελέτε για τεχνικά ζητήματα, σταθερότητα επιβατηγών πλοίων ή οχηματαγωγών. επιση λειτουργούμε δηλαδή σαν ένα είδος διεθνέ ε, consultant της Επιτροπής. Συχνά μας ζητάει η Επιτροπή να συνεργαστούμε ε, να μετάσχουμε σε διεθνείς αποστολές της ε, Επιτροπής είτε μερικές φορέ επειδή δεν έχουν το δυναμικό να αντιπροσωπεύσουμε την ε, Επιτροπή σε διεθνεί οργανισμού, όπως τον IMO, την ΙΑΛΑ κλπ. Αυτά σε ό,τι αφορά το πρώτο καθήκον. Δεύτερο καθήκον, η δεύτερη ομάδα ευθυνών που έχουμε. Μετά την, το ναυάγιο του τάγκερ του Πρεστής και την ε, τεράστια ρήπανση που προκλήθηκε, θα το θυμάστε αυτό εσείς σίγουρα κύριε Πρόεδρε, τα ευρωπαϊκά όργανα απάντησαν με ταχύτητα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα αποφασίστηκε ότι η έμψα που μόλις τότε είχε δημιουργηθεί θα έπρεπε να αναλάβει τελείως διαφορετικά καθήκοντα για να δημιουργήσει ένα δίκτυο μεγαλύτερων σκαφών μεγαλύτερου ε, δυναμικού που θα μπορούσαν να απαντήσουν ταχύτερα σε περιπτώσεις ρίσπανσης και να συμπληρώσει έτσι τα μέσα που είχαν στην διάθεσή τους τα κράτη-μέλη. Ούτως ώστε να ρουφήξουν το πετρέλαιο από την επιφάνεια πριν βουλιάξει. Είναι φθηνότερο να ε, αντλήσεις το πετρέλαιο από την επιφάνεια παρά όταν ε, θες να καθαρίσεις τις παραλίες ή τα σκάφη αργότερα. πέραν βεβαίως της ε, περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται. Στο αναμεταξύ υπάρχουν 16 τέτοια σκάφη με σύμβαση, συνήθως ΣΔΙΤ, είναι, έχουμε σκάφη που βρίσκονται στη Βαλτική, στη Βόρειο θάλασσα, στο δυτικό μέτωπο του Ατλαντικού της Ευρώπης, στη Μεσόγειο, ακόμα και στην, ε, στον Εύξηνο Πόντο. Φέτος ελπίζουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω το σύστημα με, άλλες δύο, με άλλα δύο σκάφη, με σύμβαση πάντα, για τον Βυσκαϊκό και για τον Φιλανδικό κόλπους. Έχουν ξεκινήσει 10 ε, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ε, συγγνώμη, ε, διαγωνισμού και ελπίζω το σύμβαση να ολοκληρωθεί φέτος. Επίσης έχουμε ένα σύστημα ε, ε, διαπίστωσης της ε, ρήπανσης μέσω δορυφόρου. Γιατί πέραν των μεγάλων καταστροφών που γίνονται μια φορά τα κάθε 2-3-5 χρόνια, σε καθημερινή βάση τι συμβαίνει. Πολλά πλοία που περνούν ε, που, που ταξιδεύουν τραβούν νερό για, να, νερό να καθαρίσουν τις ε, δεξαμενές τους στο πλοίο το οποίο δεν είναι νόμιμο αλλά συμβαίνει αυτές λοιπόν οι μικρές ρηπάνσεις συχνά βλάπτουν περισσότερο το περιβάλλον από ότι τα οι μεγάλες διαλογές πετρελαίου από ατυχήματα. Το σύστημα λέγεται Clean Sea Net. Λειτουργεί από τον Απρίλιο του 7 και έχει εντοπίσει εκατοντάδες τέτοιες ε, περιοχές που ρηπάνθηκαν. Υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΜΣΑ και των παράκτιων κρατών. Το σύστημα πώς λειτουργεί. 30 λεπτά μετά το πέρασμα του δορυφόρου η έκθεση με την ανάλυση βρίσκεται στο τραπέζι του κράτους που είναι αρμόδιο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Αν ο δορυφόρος διαπιστώσει ίχνη πετρελαίου, το παράκτιο κράτο είναι υποχρεωμένο να στείλει ένα σκάφο ή ένα ελικόπτερο να δει ότι πράγματι έγινε και να αναλάβει δράση κατά του ρηπαντή. Του ρηπαίνοντο, συγγνώμη και βεβαίως μπορούμε πάντα να το βελτιώσουμε, αλλά λειτουργεί και τα καλά. Η υπηρεσία Clean CNET παρέχεται στα κράτη-μέλη δωρεάν. Πληρώνεται από τον προπολογισμό της κοινότητας. Όλα τα παράκτια κράτη, καθώς και η, της Ένωσης και η Νορβηγία και η Ισλανδία μετέχουν στο σύστημα αυτό. Είναι ικανοποιημένα τα κράτη-μέλη από την υπηρεσία αυτή και το γεγονός ότι ένας οργανισμός και μόνο, η έμψα συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούσε να διαπραγματευτεί εξ όλων των παρακτήων κρατών με τις μεγάλες εταιρείες ε, δορυφόρων μας επέτρεψε να έχουμε ένα, μια καλή συμφωνία για ένα σύγχρονο σύστημα με πολύ χαμηλή τιμή. Το κεντρικό θέμα, το κεντρικό μότο του έργου της ΕΜΣΑ είναι οι οικονομίες κλίμα, κλίμακος. Μιλάμε για δορυφόρους και έτσι θα περάσω στην τρίτη ομάδα αδειοτήτων που έχει η ΕΜΣΑ. Τα συστήματα παρακολούθησης ναυτικών κινήσεων. Όσοι ήσασταν και στην προηγούμενη επίτροπη θα θυμάστε ότι τον Οκτώβριο του 2007 το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα που έλεγε ότι θα έπρεπε η ΕΜΣΑ να, παρά, να ετοιμάσει ένα σύστημα δεδομένων ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Αυτό το σύστημα ωστόσο τι σήμαινε ότι όλα τα εμπορικά σκάφη ανά τον κόσμο έπρεπε να στέλνουν τουλάχιστον τέσσερις φορές την ημέρα ε, θέση, ε, έκθεση θέσης δορυφορικά στο κράτος σημαία τους. Το οποίο πρέπει να έχει μια βάση δεδομένων αποθήκευση των μηνυμάτων αυτών και κατόπιν τα κράτη-μέλη αντικαθιστούν τις ε, εκθέσεις θέσεων για λόγους ασφάλειας. Το Συμβούλιο δηλαδή αποφάσισε ότι δεν θα δημιουργούσαν τα κράτη επιμέρους βάσει δεδομένων για το MRIT, αλλά θα ζητούσαν από την ΕΜΣΑ να ε, κάνει το σύστημα αυτό μόνο του, ακριβώς για να υπάρχουν οικονομίες ε, κλίμακας. Το σύστημα πραγματικά με περηφάνεια σας λέω λειτουργήσε, ξεκίνησε τον Ιούνιο, καλύπτει τις προσδοκίες μας, δουλεύει, μετέχουν και εκεί η Νορβηγοί και η Ισλανδία, καθώς και κάποια υπερπόντια εδάφη των κρατών μελών. Το, η βάση δεδομένων ή της Ένωσης MRIT καλύπτει 30% του των χωρών του κόσμου και 25% του στόλου, του παγκόσμιου στόλου. Ξέρουμε λοιπόν που βρίσκονται τα σκάφη μας, όπου και να βρίσκονται. Τελειώνοντας. Αλλά πάντα για το LRIT. Αυτό που θέλαμε να δούμε είναι κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να βοηθήσουν την αντιμετώπιση της πειρατείας. Επικοινωνήσαμε την UNAFOR και την επιχείρηση Αταλάντη που έδειξαν ενδιαφέρον. Εν ολίγης, από τις 25 Σεπτεμβρίου παρέχουμε πληροφορίες LRI, θέσεων LRIT στην UNAFOR αλλά μόνο για τα πλοία κρατών της Ένωσης που επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Αυτό επιτρέπει καλύτερη οργάνωση της προστασίας και και πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων που υπάρχουν. Τώρα, ε, πώς, τι γίνεται με την ε, παρακολούθηση των, της κίνησης των σκαφών στα δικά μας ε, χωρικά είδωτα. Θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω ένα σύστημα που λέγεται Safe για να παρακολουθούμε την κίνηση των σκαφών με μεγαλύτερες λεπτομέρειες στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα. Το σύστημα επιτρέπει να έχουμε και πληροφορίες για το φορτίο αν υπάρξει ατύχημα, ξέρω, ένα κάποιο πρόβλημα με το σκάφος. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τις πληροφορίες αυτές γρήγορα. Σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, το σύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί σε μία περίοδο 5 ετών και άρχισε να λειτουργεί και αυτό το καλοκαίρι. Βρισκόμαστε σε μία φάση ε, ρονταρίσματος προσπαθώντας να το συνδέσουμε με, τα, με τις υπηρεσίες των κρατών μελών. Θα έχει πάνω από 2.000 εγκεκριμένους χρήστες, 1.000 λιμάνια, κέντρα διάσωσης στη θάλασσα, όλες τις υπηρεσίες ε, που χρειάζεται να έχουν εικόνα. Το SafeCNet θα είναι η σπονδυλική στήλη όλων των ε, συστημάτων ενημέρωσης για την αυσιπλοεία. Τώρα, ποιε είναι οι προοπτικές για το μέλλον. Το επόμενο βήμα είναι να ενοποιήσουμε όλα τα συστήματα παρακολούθησης της κυκλοφορίας της, ε, στην θάλασσα, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό και νέα προϊόντα. Παράδειγμα, αν συνδέσεις το CleanSynet και το SafeSynet, θα έχεις εικόνα όχι μόνο των ιχνών πετρελαίου, αλλά και την ταυτότητα του σκάφους που ρηπαίνει τη θάλασσα. Θα εντοπίσεις στην οθόνη σου τον ρηπαίνοντα. Αυτό στο στόχο τον έχουμε για το 2010. Δεύτερο θέμα. Το σύστημα αυτό παρακολούθησης της ναυσιπλοείας με δορυφόρου μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλους, τη Frontex για παράδειγμα, που έχουν την ευθύνη της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Δεν είναι δική μας δουλειά, αλλά για τους στόχους τους και αυτοί θέλουν να έχουν ένα σύστημα παρακολούθησης της κίνησης στη θάλασσα. Ιδίως στα εξωτερικά σύνορα, στα θαλάσσια εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Σε συνεργασία με την υπηρεσία επαφών εξετάζουμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε. Το ίδιο και με την υπηρεσία, ε, με τον οργανισμό αλίας. Και αυτοί θέλουν να έχουν έλεγχο των αλληλευτικών σκαφών που βρίσκονται, τι κάνουν. Υπογράψαμε μια συμφωνία για να διερευνήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί και με αυτούς. Σας είπα για τη UNAFOR, για την επιχείρηση ταλάντη αυτές τις μέρες μας επισκέπτονται και κάτι ναύαρχοι για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η Επιτροπή βεβαίως είναι αυτή από όπου προήλθαν οι προτάσεις αυτές. Εξετάζει την δυνατότητα πολλαπλής χρήσης των συστημάτων πληροφόρησης ε, από πολλούς οργανισμούς στην Ένωση. Επίσης, η Επιτροπή ξεκίνησε την ιδέα της στενότερης συνεργασίας με την πολιτική γειτονία, μέσω της πολιτικής γειτονίας με τις ε, Γειτονικέ χώρε. Ο αντιπρόεδρο κ. Σταγιάννη αναφέρθηκε σαφώς για το θέμα αυτό. Θα ήθελε η ΕΜΣΑ να εμπλέκεται περισσότερα στην ε, ε, συνεργασία με τις χώρες της βορειο αυτική, στον τομέα της θαλάσσιας της ασφάλειας στην αυσιπλοεία και της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα μέλη της Επιτροπής, Πρόεδρε, ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα σταματήσω εδώ. Πολλά κάναμε τα τελευταία έξι χρόνια, πολλά μένουν να κάνουμε. Ελπίζω να μας επισκεφτείτε λοιπόν μια μέρα στη Λισαβόνα και να δείτε τους 200 περίπου υπαλλήλους που με πάθος δουλεύουν για, την, για το έργο μας το καινούριο μας κτίριο, πανέμορφο κτίριο. Είμαι, θα είμαστε περήφανοι να σας δείξουμε σε τι χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά και οι οδηγίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντερόιτ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ξετυλίγεται το κουβάρι της Έρικα. Θα περάσουμε πρώτα στους συντονιστές, τρία λεπτά, μετά τα μέλη δύο λεπτά, συνολικά 30 λεπτά. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιστοί στη διαδικασία. Κύριε Σκουίνα από το ΕΛΚ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και την εργασία που κάνει η ΕΜΖΑ σε σχέση με την ασφάλεια των πλοίων αλλά και της θάλασσας τη δουλειά που κάνει για μας ε, και για τα κράτη-μέλη. Είναι μεγάλη σημασία, ειδικότερα όσον αφορά και στην ρήπανση των θαλασσών. Με μεγάλη προσοχή παρακολουθήσαμε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ασχολείστε και με την εκπαίδευση των ναυτικών. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει προσωπικό από τρίτε χώρες ε, που είναι καλά εκπαιδευμένο, πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένο γιατί ταξιδεύει στις θάλασσές μας, ε, στον Βυσκαϊκό, στην Μεσόγειο και στη Βόρειο Θάλασσα. Οι τεχνικές ε, προδιαγραφές επίσης για την ασφαλή χρήση των πλοίων είναι ένα άλλο θέμα και τη λειτουργία τους διότι υπάρχει και μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων και από κοινού ε, έχουμε αποφασίσει να μην έχουμε ε, πλέον ε, πλοία μονοκίτους για οικολογικούς λόγους και το σύστημα που έχω έχετε φτιάξει, το Clean Net, επίσης είναι πολύ σημαντικό. Η συνεργασία μεταξύ του οργανισμού σας και των αρχών και εθνικών κρατών είναι φυσικά, ε, παίζει φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο. Και αν καταφέρουμε να παρακολουθήσουμε όχι μόνο τις ιδιαίτερα επικίνδυνες μεταφορές πετρελαίου ή επικίνδυνων προϊόντων, αλλά να δούμε και τις ε, περιβαλλοντικές αμαρτίες ε, που ρηπαίνουν τα ύδατά μας μέσω δορυφόρων και σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές που ε, χρησιμοποιούν ας πούμε ε, τα, αεροπλάνα τους, ας πούμε στη Γερμανία έχουμε 128 αισθητήρε ε, πετρελαίου, τότε θα έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Επίσης, ε, σημαντικό ρόλο παίζει το πώς το Γαλιλαίο, το σύστημα αναυσιπολογίας ε, θα συμπεριληφθεί σε αυτήν την διαδικασία προστασίας. Όλα αυτά παίζουν πολύ αποφασιστικό ρόλο θα έλεγα όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα. Ήδη βλέπω τον πρόεδρο να μου λέει να σταματήσω. Εδώ Επίσης να πω ότι είναι σημαντικό να συντονιστούμε με την ΕΜΖΑ έτσι ώστε να δούμε πώς ε, θα συντονίσουμε τις δυνάμεις μας σε περίπτωση που βρίσκεται σε κίνδυνο ένα πλοίο ε, στη θάλασσα. Πρέπει να βρούμε δυνατότητες ρημούλκησης οι οποίες θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Και αυτό θα πρέπει ε, στο μέλλον να γίνεται πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κιούν που αναγνωρίζει τους περιορισμούς ε, χρόνων, ο κύριος Αλκαντρουή από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Ντερούιτ ε, για την πολύ ε, ξεκάθαρη παρουσίαση. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, όπως είπε ο κύριος Κιούν, η ρήπανση από τα πλοία που καθαρίζουν τις δεξαμενές τους και τα λοιπά, υποδιάζουν τις δεξαμενές τους. Χρησιμο... Αναφερθήκατε στη χρήση τεχνολογίας ε, που χρησιμοποιείται για να γίνει αυτό. Ε, βλέπετε κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά των ε, πλοίων όσον αφορά αυτό το θέμα. Πόσους ρηπαίνοντες πιάνουμε επαυτοφόρο κάνοντας, χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα. Κοίταξα το φυλάδιό σας, δεύτερη ερώτηση. Στη σελίδα 3 υπάρχουν κάποιες στατιστικές που αφορούν κάποια από τα ατυχήματα που έχουν αναφερθεί μεταξύ 2004-2008. Υπήρξε σχεδόν διπλασιασμός ε, των ε, ατυχημάτων. Βέβαια δεν λέγεται πόσο σοβαρά ήταν τα ατυχήματα. Αυτό οφείλεται στην καλύτερη αναφορά των ατυχημάτων, ε, χειρότερη χρήση των πλοίων ή σε άλλες αιτίες. Και τελευταία ερώτηση, είπατε ότι σε κάποιες περιπτώσεις εκπροσωπείται την Επιτροπή. Για παράδειγμα στον ε, IMO, το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, οπότε αναρωτιέμαι εν ώψη και της διάσκεψης της Κοπενχάγης. Ξέρουμε ότι χρειάζονται πολλά να γίνουν για το καθαρισμό της ε, ναυσιπλοείας και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε σε διεθνές επίπεδο, να μειώσουμε ειδικότερα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Να μας πείτε λοιπόν μερικά πράγματα σχετικά με το πώς έχουν ε, τα πράγματα ως τώρα. Δύο λεπτά και 55 δευτερόλεπτα χρησιμοποίησατε. Μπράβο. Ε, από την ομάδα ALDE, κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ για αυτή την εξαίρετη παρουσίαση που μας ε, δίνει τόσες δυνατότητες για συμπεράσματα. Έχω δύο ερωτήσεις. Ε, θα είμαι κάτω από τρία λεπτά. Η πρώτη έχει να κάνει με τα συστήματα δορυφόρων. Είπατε ότι σε αυτά τα συστήματα δεν έχουν όλα τα κράτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ε, σημαία τους. 35 ε, είναι τα κράτη. Θα έπρεπε να έχουμε, νομίζετε εσείς, όλα τα κράτη σε αυτό. Και πώς θα το κάνουμε. Δεύτερη ερώτηση. Όταν έχουμε ε, τους δορυφόρους δεν έχουμε μόνο στοιχεία για το πετρέλαιο αλλά και άλλες μορφές δεδομένων. Ε, διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε μόνο τα στοιχεία που και μεταδίδουμε τα στοιχεία που αφορούν στην ε, ρήπανση λόγω πετρελαίου και τα και όχι άλλα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μάισνερ για τους πράσινος, ο κύριος Κράμερ φυσικός. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το Clean Sinet ιδιαίτερα. Συχνά ε, αναφέρεται ότι υπάρχει ένα παιχνιδάκι μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και IMO. Όταν ήταν εδώ ο κύριος Πίτσικε, εγώ δεν ήμουν εδώ, είπε ότι υπάρχουν στον IMO κανόνες ε, που εφαρμόζονται μόνο από τρία ή τέσσερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το επιβεβαιώνεται. Και τι γίνεται όταν δεν περνάνε οι κανόνες του IMO στα εθνικά δίκαια. Μετά τι γίνεται όταν έχουμε ένα ε, πλοίο σε ένα λιμάνι που ρηπαίνει τα νερά. Όταν μέσα από το σύστημα ε, δορυφόρου ανακαλύπτεται ένα τέτοιο πλοίο, τι γίνεται, πόσο υψηλά είναι τα πρόστιμα. Είναι τόσο ψηλά όσο να πραγματικά να τους παραδειγματίζουν. Και το τελευταίο θέμα, το είπα και η κυρία Μάισνερ, μπορεί να υπάρξει μια άδεια ε, στα ύδατα των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ταξιδεύουν ε, μόνο πλοία τα οποία θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Επίσης, ε, με την αεροπορία ε, έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε το ίδιο, να μην υπάρχουν εξαιρέσεις δηλαδή στα αεροπλάνα που τηρούν τους κανόνες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βαντάμ για το ίσιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ντεράιτο. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Έχω δύο ερωτήσεις. Μία διαδικαστική και μία της ουσίας. Όσον αφορά τα διαδικαστικά, όπως και με άλλες υπηρεσίες έχουμε το ίδιο πρόβλημα και εδώ. Οι θέσεις που κατέχουν, δηλαδή πρέπει να δικαιολογούν τη δουλειά που κάνουν. Ξέρω ότι είσαστε σύμβουλος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσατε όμως να μου πείτε σε ποιον είσαστε υπόλογος όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ποιος σας ελέγχει. Θα ήθελα ακριβή απάντηση. Αναφερθήκατε σε ομάδες επιθεώρησης που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Ξέρω ότι όσον αφορά την εσωτερική ναυσιπλοεία υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά ε, αγαθά που έρχονται από την Κίνα. Ε, μπορείτε να μας πείτε. για τις ασφαλίσεις όσον αφορά την κάλυψη, την ασφαλιστική που υπάρχει στην Κίνα όσον αφορά τα σκάφη αυτά που έρχονται στην Ευρώπη. Μήπως υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα, υπάρχει με την εσωτερική ναυσιπλοεία και με τις κανονικές θαλάσσιες μεταφορές. Κύριε Ντερόιτερ, έχετε κάποιες ερωτήσεις αν μπορείτε να είσαστε πειθαρχημένοι όσον αφορά το χρόνο. Ένα δεκάλεπτο για να απαντήσετε και έτσι έχουμε το χρόνο και να απαντήσουν και τα μέλη. Well, thank you for... Uh, Ευχαριστώ για τις πολύ εμπνευσμένε ε, ερωτήσεις σας. Σας προσπαθήσω να απαντήσω με ξεκάθαρο και συνοπτικό τρόπο. Πρώτον, πώς μπορεί η ΕΜΣΑ να βοηθήσει καλύτερα τα παράκτια κράτη τα οποία αντιμετωπίζουν εκτακτής, περιπτώσεις εκτακτής ανάγκης και ατυχήματα. Ερώτηση του κυρίου Κούν. Να υπογραμμίσω ότι η ΕΜΣΑ δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Η, το Τα καθήκοντα της ακτοφυλακής ε, υπόκεινται στα κρατημέλη. Αυτά είναι που ε, ορίζουν τι γίνεται στα χωρικά του ύδατα. Η ΕΜΖΑ δίνει κοινά και καλύτερα εργαλεία ώστε οι ακτοφυλακές να έχουν καλύτερες πληροφορίες και πιο γρήγορες και έγκαιρες πληροφορίες ε, μέσα από το Safe για το τι κάργο, τι φορτίο μεταφέρεται. Δεν το ανέφερα, αλλά έχουμε και ένα σύστημα για τις χημικές ουσίες αν υπάρχει ένα χημικό τάνκερ, το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αν βρούμε τη χημική ουσία, ε, η εκτοφυλακή δεν γνωρίζει τις ιδιότητες. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα με την, μέσω της Ευρωπαϊκής Χημικής Βιομηχανίας που ε, δίνει τη δυνατότητα στην ακτοφυλακή να έχει σύνδεση με την ε, εταιρεία που φτιάχνει την ουσία έτσι ώστε να τους δίνει συμβουλές για το τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Είναι λοιπόν επιπλέον εργανηλία για τη σωστή ε, λειτουργία και την αντίδραση, τη σωστή αντίδραση στην ρήπανση. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις για το Clean Sinet και αυτό είναι κατανοητό, γιατί είναι ένα σύστημα που πάντοτε τραβά την προσοχή. Πόσες διώξεις με βάση του, το Clean Sinet, αυτή ήταν μια ερώτηση. Αυτό το σημείο πραγματικά χρήζει περαιτέρω προσοχής υπάρχει μια σειρά κρατών μελών που έχουν ε, οργανώσει πολύ αποτελεσματικά τις διώξεις. Δεν θέλω να αναφέρω κράτη-μέλη, αλλά να πω ότι ο δημόσιος κατήγορος στην Πρέστε, στη Γαλλία, είναι ειδικό στην αυσιπλοεία και δεν διστάζει. Μόλις βρεθεί ένα πλοίο μέσω του δορυφόρου πηγαίνει ένα αεροπλάνο του ναυτικού και επικυρώνει ότι αυτό είναι το πλοίο, αυτό είναι πετρέλαιο και αυτό αρκεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της δίωξης. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει επιτύχει πρόστιμα και πραγματικά ε, τα τα πρόστιμα είναι πολύ ψηλά, 400-500 ευρώ. Επίσης έχουμε δει περιπτώσεις όπου ο δορυφόρος βρήκε τον ρηπαίνοντα, το πλοίο πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο λιμάνι της περιοχής ε, και ε, δεν τους ε, συλλάβαμε, αλλά τέλος πάντων τους υποχρεώσαμε να πληρώσουν. Η δίωξη βέβαια οργανώνεται διαφορετικά σε κάθε κράτος μέλος σε κάποιες δικαιοδοσίες χρειάζονται περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία. Ποιος ήταν αυτός ε, που έδωσε την εντολή, ας πούμε, για να ανοίξουν τα πάρια είναι κάτι που θέλουν να ξέρουν. Και αυτό ε, δυσκολεύει την επιτυχία της δίωξης. Δεν είναι δουλειά της ΕΜΣΑ αυτό. Εμείς ε, απλώς δίνουμε τα εργαλεία για να ταυτοποιηθούν οι πιθανοί ρηπαίνοντες και η ρήπανση. Θα ήθελα όμως να ανοίξει η συζήτηση μεταξύ των διοκτικών αρχών ε, στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να μιλήσω με την Κομισιόν. Δεν είναι βέβαια στο, στη δική μας εντολή, αλλά πρέπει αυτά τα μέρη να, έλθουν, να συνέλθουν και να συζητήσουν για να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Μια άλλη ερώτηση είχε να κάνει με την αύξηση των ε, περιστατικών ε, ε, στην περίοδο 2004-2008. Δεν ξέρω αν θα είναι επιστημονική απάντησή μου, δεν υπάρχει μάλλον, αλλά τότε ήταν η χρονιά της έξαρσης τεράστια ε, χρήση ε, πλοίων και μεταφορών. Ήταν δύσκολο να βρούμε κατάλληλο προσωπικό, οπότε στο διάστημα 2004-2008 υπήρξαν πολλά ατυχήματα λόγω ανθρωπίνου λάθους. προβλήματα με τις μηχανές, γιατί δεν υπήρχε κανείς στο μηχανοστάσιο, ήταν όλα πλήρως αυτοματοποιημένα. σαράξεις κτλ. Τώρα ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μείωση. Δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον δεν έγινε ε, κάποια τεράστια καταστροφή. Υπήρχαν επίσης κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να το συνδέσω αυτό και με το θείο. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πεδίο. Έχουν γίνει πολλά στην Ευρώπη για τη μείωση των εκπομπών από τα αυτοκίνητα, τα τρένα, από τις ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού. Όμως η ναυσιπλοεία έχει ξεφύγει γιατί δεν αφορά μόνο τον Ευρωπαίο νομοθέτη αλλά ε, τη διεθνή αγορά και ο ΑΕΛΟ ήταν πολύ αργός ως προς αυτό. Ο ΑΕΜΟ όλο και περισσότερο πιέζει, έχουν υιοθετηθεί κάποια μέτρα, αλλά ο χρόνος εφαρμογής ε, μάλλον είναι βραδύς. Για τη Βόρεια Ευρώπη έχει οριστεί ένας ε, χώρος ε, ε, ελέγχου των εκπομπών και υπάρχουν πιο φιλόδοξα στάνταρ. Μιλάμε και για τη ρήπανση θείου λόγω των πλοίων, γιατί τα καύσιμα των πλοίων υπάρχουν περιέχουν πολύ θείο. Είναι περίεργος ο μηχανισμός. Όσο πιο καθαρά καύσιμα απαιτούμε στη γη, τόσο περισσότερο θείο και άλλα ε, ρηπαντικά στοιχεία ε, ως υπολείμματα ε, καυσίμων έχουμε από τα πλοία. Δεν θα μπω σε πιο επιστημονικές λεπτομέρειες. Υπάρχουν οι διάφορες υπηρεσίες της Κομισιόν που ασχολούνται με την πολιτική γι' αυτά. Επίσης, υπήρξε μια ερώτηση από την κυρία Μάισνερ για την πειρατεία. Να πω ότι όλα αυτά είναι πολύ πρόσφατα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μόλις πριν από δύο εβδομάδες, στείλαμε ένα μήνυμα σε όλα τα κράτη-μέλη και είπαμε ότι μπορούμε πλέον από τεχνική άποψη να δώσουμε πληροφορίες στη UNAFOR αν μας δώσετε την άδεια. Μια σειρά κρατών μελών άμεσα απάντησαν μέσα σε μία μέρα, μέσα σε δύο μέρες. Υπάρχουν λοιπόν πέντε κράτη, δίνουμε στοιχεία στο στρατό και είμαι σίγουρος ότι μετά από λίγο χρόνο σκέψης όλα τα κράτη θα δώσουν την αδειά τους. Αυτό ελπίζω τουλάχιστον. Εμείς συζητούμε ε, ατομικά με το κάθε κράτος. Η προστασία των δεδομένων, άλλη μία ανησυχία. Το σύστημα ε, είναι κλειστό μεταξύ της ΕΜΖΑ και εγκεκριμένων χρηστών. Για το CleanSynet δεν είναι πρόβλημα γιατί υπάρχει μικρός αριθμός χρηστών. Για το SafeSynet υπάρχουν πάνω από 2.000 εγκεκριμένοι χρήστες. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι αυτοί πειθαρχημένοι. Να μην ε, αποκαλύπτουν στοιχεία σε μία εγκεκριμένα μέρη. Γιατί ε, πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι ευαίσθητες. Η σχέση μεταξύ του IMO, της θέσπισης κανόνων και της θέσπισης κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν συνήθως ε, μεταφράζει όλους τους σχετικούς κανόνες του IMO σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχει ξεφύγει κάτι μίζωνος σημασίας. Ε, οι περισσότεροι κανόνες ε, μεταφέρονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πολλές φορές με συγκεκριμένες προσθήκες. Υπήρξε και μία ερώτηση από τον κύριο Κράμερ για το Μάρπολ, για την σύμβαση σχετικά με τη ρήπανση. Η Μάρπολ επιτρέπει την άντληση ελάχιστες ποσότητας ε, πετρελαίου στην ανοιχτή θάλασσα, όχι στα παράκτια ύδατα. Και συγκεκριμένα ορίζεται τι μπορεί να κάνει κανείς στη μέση του ωκεανού και τι στα παράκτια ύδατα. Με λίγα λόγια, αυτό σημαίνει στις παράκτιες περιοχές ε, των ζωνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν μπορείς ε, να ρίξεις στο νερό κάτι που έχει ορατό ε, πετρέλαιο. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο το σύστημα και πραγματικά ανοιχνεύει ακόμα και πολύ μικρές ποσότητες πετρελαίου. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις, γιατί δεν έχω χρόνο. Α, ναι, έχω την πιο ε, δύσκολη ερώτηση. Για την τιμωρία δεν είπατε αν τους ανακαλύψουμε. Μάικ, από τον πρόεδρο οι επισημάνσεις. Θα, γινόταν, θα είχαμε αναρχία να το κάναν όλοι αυτό. Το επίπεδο των κυρώσεων. Αυτό το κρίνει ο δικαστής. Αυτή είναι η βασική αρχή. Εδώ όμως υιοθετήσατε κάποιους κανόνες για ποινικέ κυρώσεις όσον αφορά τη ρήπανση που προξενείται από σκάφη. Οι κυρώσει δεν είναι εναρμονισμένες, αλλά προβλέπει ο νόμος ότι οι υπεύθυνοι για τη ρήπανση από πλευρά σκαφών, ρήπανση θάλασσα από πλευρά σκαφών, μπορούν να τιμωρηθούν όχι μόνο μέσω διοικητικών ποινών και προστήμων, αλλά και ποινικέ κυρώσεις μπορεί να επιβληθούν. Και αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Ε, ο, ο που δίνει εντολή στον πλοίαρχο να αδειάσει πετρέλαιο στη θάλασσα μπορεί θεωρητικά να καταλήξει στη φυλακή. Θα ήθελα να είμαι αρκετά γενναίος για να απαντήσω στο ερώτημα του Πέτερ Βαντάλεν. Σε ποιον είστε υπόλογος, ήταν το ερώτημα. Σε ποιον λογοδοτείτε. Το αφεντικό μου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της υπηρεσίας μας. Εκεί εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολυπληθή αντιπροσωπεία. Και είναι ο που διορίζει το διευθυντή της υπηρεσίας που εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας, που μπορεί να απολύσει το διευθυντή, να απορρίψει το πρόγραμμα εργασίας, τον προπολογισμό, την ετήσια έκθεση και όλα αυτά. Πέραν αυτού όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλεί τους διευθυντές των υπηρεσιών και πρέπει να έρθουμε και να εξηγήσουμε τι κάνουμε με τον προϋπολογισμό που ε, μας δώσατε. Το Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις τεχνικής φύσεως και το κάνει το Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Μεταφόρων, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει όλες τις δραστηριότητες της υπηρεσίας κάθε χρόνο δεχόμαστε επίσκεψη που κρατά αρκετέ εβδομάδες δεν αφήνουν λίθον επί Γυρίζουν κάθε λιθαράκι και ψάχνουν. Άρα υπάρχει κάποιος έλεγχος. Και έτσι έπρεπε να είναι άλλωστε. Και τέλος και το θέμα της ποιότητας της χαλιβουργίας στην Κίνα ήταν το ερώτημα. Και ήταν θέμα στις θαλάσσιες μεταφορές την εποχή της ακμής 2006-2007. Οι πλειοκτήτες παράγγελναν τόσα πολλά καινούργια σκάφη, κάτι που το έχουμε μετανιώσει τώρα, που κάθε ε, ε χαλιβουργείο στην Κίνα αυτό το ε, ναυπηγείο. Είχαν ε, γεμάτο το πελατολόγιο τους επί τρία χρόνια. κατασκεύαζαν ακόμα και στόχους των ποταμών ε, να φυγούσαν πλοία. Όπου υπήρχε ανοιχτός χώρος. Ασχολιόταν περισσότερο με σκάφη εσωτερική ναυσιπλοεία παρά με τα μεγάλα ποντοπόρα σκάφη. Ε, λόγω δυνατότητας της βιομηχανία. Γι' αυτό οι νιογνώμονε έπρεπε να συμμετάσχουν στο παιχνίδι, να μπορέσουμε να πιέσουμε όσον αφορά την ποιότητα της κατασκευής. Αλλά λόγω της άνθησης στην αυπηγική ε, είχαν πρόβλημα έλλειψη προσωπικού οι νιογνώμονες για να ελέγχουν τα σκάφη. Αλλά εμείς ήμασταν αρκετά αυστηροί. Δεν νομίζω ε, κάπου να υπάρχει κάποια ορολογιακή βόμβα που απειλεί ε, τα νέα σκάφη Δηλαδή να έχουμε νέα σκάφη ποντοπόρα τα οποία δεν πληρούν τι προδιαγραφέ τι ποιοτικέ. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα σα έκοβα εδώ, λέει ο Πρόεδρο, γιατί έχουμε μείνει πίσω χρονικά και έχουμε και άλλου που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσει. Έχουμε και του 10 συντονιστέ που περιμένουν. Αλλά είναι σωστό αυτοί που είναι γεγραμμένοι να πάρουν το λόγο. Δεν θα βάλω κι άλλον στο κατάλογο όμω. Ε. Ο κύριος Μπλάστο είναι επόμενο. Η κυρία Μπλάστο, διορθώνει ο Πρόεδρο. Μπιλμπάρ, Γκράντες Πασκάλ, Κάλτσιν κλπ. Και μετά τέρμα, γιατί θα ξημερωθούμε εδώ. Η ε, κυρία Βλαστό, ένα λεπτάκι, ε. θα σα ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα προχωρήσω και τα γρήγορα. Κύριε Διευθυντά, αναφερθήκατε στην επιθεώρηση των σκαφών και στην προηγούμενη θητεία είχα τη χαρά να είμαι συγκήτρια πάνω στο κείμενο που αφορά τον έλεγχο από το κράτος λιμένος. Το κείμενο θέλει ενισχύσει τις επιθεωρήσεις των σκαφών και στα λιμάνια ε, και στις δεξαμενές. Αρκετά σημαντική βάση δεδομένων απαιτείται για αυτόν τον σκοπό και προτείναμε να υπάρξει ένα νέο σύστημα επιθεωρήσεων και ελέγχων για κάθε σκάφος θα μπορούμε να διαπιστώνουμε αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος και τους ελέγχους ότι ενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θαλασσίων ε, Μεταφορών, Θαλασσίας Ασφάλειας, Ασφαλείας μάλλον Θαλασσίων Μεταφορών. Έχουμε βάση δεδομένων, θα ξέρουμε κάθε σκάφος από τι κινδυνεύει, ποιο είναι το ιστορικό των ε, επιθεωρήσεων. Εσεί θα δημιουργήσετε τη βάση δεδομένων, έτσι. Και η υπηρεσία έχει δημιουργήσει ένα σύστημα. Το ΦΕΤΙΣ 2 e έχει δημιουργήσει και θα συνδέεται και με άλλη βάση δεδομένων. Το CFSINET και θα είναι προσβάσιμο από τα κράτη-μέλη του Μνημονίου των Παρισίων. Κύριε Διευθυντά, μπορείτε να μας πείτε πώς προχωράει η όλη ιστορία, πότε θα λειτουργεί και το θέτης θα είναι βάση πληροφορικής και τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στο υπόμνημα των Παρισίων θα βρίσκουν τις ε, πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη τους και με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει το κάθε σκάφο. Κύριε Μπεμπάου, για ένα λεπτό και πάλι, μα σας παρακαλώ, θα ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Ντερόιτερ για τι εξηγήσεις που μας έδωσε. Συγκεκριμένε ερωτήσει θέλω να θέσει. Δύο μίλησε για τα σκάφη που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την, την ρήπανση και για το ότι είχε 16 σκάφη που ε, έχουν καθώς και ότι στο τέλος του έτους θα, μας, θα έχουν άλλα δύο σκάφη, ένα από τα οποία θα είναι στο Βυσκαϊκό κόλπο. Πού ακριβώς. Δεύτερον, ποιο είναι το κόστος της ε, συνδρομής των 16 αυτών σκαφών και τη συμπερίληψη στο τέλος του έτους άλλων δύο όπως αναφέρατε και ποιο είναι ο αριθμός των επεμβάσεων που έχουν πραγματοποιήσει. Επίσης, σε ό,τι αφορά την επιχείρηση Αταλάντη, Δυστυχώ, κατήγγειλα στο Κοινοβούλιο σε δύο ευκαιρίε, την έλλειψη προστασίας των αλευτικών σκαφών. Ένα σκάφος αυτές τις μέρες έχει ε, υποστεί πειρατεία το Αλακράνα από την περιοχή μου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σκάφο, αυτό το σύστημα RALIT ε, και θέλω να ξέρω κατά πόσον το, το Ισπανικό κράτος ζήτησε τη συνδρομή σας για την υλοποίηση, την εφαρμογή του συστήματος αυτού στην αναζήτηση των δικών του σκαφών. Ευχαριστώ. Κύριος Πασκουάλ. Ευχαριστώ. Κύριε Ντερόιτερ, εδώ όπως ξέρετε παρακολουθούμε την πορεία της, ε, του οργανισμού σας. Ήμουν ε, ιδιαίτερα, είχα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για, τη δική σας, ε, για το δικό σας οργανισμό. Ήμουν και εισηγητής κλπ. Στη δουλειά που έκανα είπατε ότι οι ερωτήσει μου είναι εξή. Πρώτον, τη ίδια με αυτή της κυρίας Μπιλμπάου. Το νέο σκάφος στο βυσκαϊκό κόλπο, πού θα λειτουργεί, τι εμβέλεια θα έχει, πότε προβλέπεται να υλοποιηθεί η συμφωνία, η σύμβαση αυτή. Δεύτερον, είπατε ότι προσφέρετε τις υπηρεσίες σας για την καταπολέμηση της πειρατείας και ότι κάποια κράτη είπαν ναι και κάποια άλλοι που δεν έχουν πει τίποτα. Η ερώτησή μου είναι, ε, δέχθηκε προσφέρατε την, την ε, ενημέρωση αυτή στην Ισπανία, το δέχθηκε. Και επίση πόσο, σε τι βαθμό τελειοποίησης έχει φτάσει το σύστημα της ε, διερεύνησης ε, των, της ρήπανης από σκάφη. Υπάρχει δυνατότητα ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση υπετιότητας ή ε, βαριάς αμέλειας. Το σύστημα μπορεί να βεβαιώσει απόλυτα την διάκριση μεταξύ ελαφράς και βαρίας αμέλειας τους ώστε να εμφανιστούν και ποινικές χειρώσεις κατόπιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Γρήγορα. Γρήγορα θα ήθελα να συγκρατήσω από αυτά που είπατε ότι στο μέλλον θέλετε να εμβαθύνετε όλο και περισσότερο στο ελοκληρωμένο σύστημα. Αναφερθήκατε στις ενδεχόμενες συμφωνίες που έχουν δρομολογηθεί με το Frontex. Όπως ξέρετε, όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αυτή η δουλειά σας, η συνεργασία με τη Frontex, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το υπογραμμίσω. Και επειδή αυτή η δραματική κατάσταση θα πρέπει να βρει λύση το ταχύτερο δυνατό και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και με τον έλεγχο που επιβάλλατε και με αυτή τη συμφωνία αυτή η συμφωνία μας στο μέλλον πρέπει να είναι, θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαι εδώ για πρώτη φορά και ακούω διάφορες υπηρεσίες που υπάρχουν. Βασική τους, ε, βασική τους μέρημνα είναι να λειτουργούν ορθολογικά. Το ολοκληρωμένο σύστημα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και των ομόρων χωρών. Το υπογράμμισε αυτό επίτροπός μας και είναι πολύ σημαντικό για να λειτουργήσει σωστά αυτή η στρατηγική που αναφέρατε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και είμαι ευγνώμων στα μέλη που είναι πολύ σύντομα. Ο κ. Χούιας έχει το λόγο. Ο κ. Αουτζίας. Λοιπόν, λέει ο κ. Αουτζίας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο, συντομότατος, λακωνικός, επιγραμματικός προς την πρόληψη κινείται η υπηρεσία περισσότερο παρά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ρήπανσης αφού συμβούν. Κανονιστικά, νομικά, ποια είναι τα προβλήματα. Αυτά που έθιξε και προηγουμένως ο κ. Κράμερ όσον αφορά αρμοδιότητες, ε, κυρώσεις, νομολογία. Τι προβλήματα τέτοια αντιμετωπίζει η υπηρεσία σας. Και θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποια θέματα που οδηγούν ίσως στην έννοια του ευρωπαϊκού υδάτινου χώρου. Υπάρχουν τέτοιες ζώνες όπως μεταξύ Κορσικής και Σαρδινίας. Ε, υπάρχει χώρος όπου μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας έχει συναυθεί σύμβαση για, την, για τον έλεγχο της μετακίνησης επικινδύνων φορτίων. Η υπηρεσία θέλει νέα μέσα ούτως ώστε και άλλες χώρες μέλη να ελέγξουν επικίνδυνες δραστηριότητε σε παρεμφερείς ε, χώρους υδάτινους όπως αυτός. Ευχαριστώ κύριε Όγκιας. Ο κύριος Ντερόιτερ ας απαντήσει σου σύντομα γίνεται και αν δεν απαντήσετε τώρα προφορικά σε όλα τα ερωτήματα μπορείτε να στείλετε, να δώσετε κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να έρθετε σε επαφή με τα μέλη να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για τον έλεγχο για τη βάση δεδομένων της χώρας λιμένος θα λειτουργεί το σύστημα μέχρι την 1η Πρώτου 2011. Το πρόγραμμα προχωράει καλά και συνεργάζονται όλα τα κράτη-μέλη. Η κυρία Μπιλμπάου και ο κ. Γκάντε Πασκάλ έθεσαν ερωτήματα. Τα νέα σκάφη για φέτο. Θα είναι στο Βυσκαϊκό κόλπο και στον κόλπο της Φινλανδίας. Ε, έχει δημοσιευτεί διαγωνισμός και καλούμε ιδιωτικούς φορείς, πλειοκτήτες να υποβάλουν προσφορές. Δεν ξέρω πού θα βρίσκονται τα σκάφη, πού θα βρίσκεται το σκάφος. Απλώς αναφέραμε το πού θα έπρεπε σε ποια περιοχή. Το κόστος δεν είναι μεγάλο. Το σύστημα έχει περίπου 22 εκατομμύρια προπολογισμό το χρόνο για την ε, αντιμετώπιση του, της ρήπανση. Είναι δορυφορικό το σύστημα που χρησιμοποιείται, το Cleansing Net και καλύπτεται το όλο σύστημα από αυτό το προπολογισμό που προανέφερα. Έχει γίνει παρέμβαση έχουν κληθεί αυτά τα σκάφη τρεις φορές να κινηθούν, να δράσουν στην Ισπανία. Η επιχείρηση Αταλάντα κατά της πειρατείας, αν απάντησε ήδη η Ισπανία, δεν ξέρω απ' έξω, πρέπει να το ελέγξω. Πιστεύω ότι θα υπάρξει υποστήριξη της όλης ε, ενίας, της όλης ιδέας. Το cleansing net μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ επιπέδων αμελίας. Όχι είναι η απάντηση. Βέβαια ο δορυφόρος δίνει κάποιες ενδείξεις αν η κοιλίδα είναι μεγάλη ή μικρή. Αλλά η παλήθευση γίνεται από αεροσκάφη και ελικόπτερα. Επιτόπια διαπίστωση και αυτό είναι που έχει σημασία για την δημιουργία της δικογραφίας. Τώρα, συνεργασία με τη Frontex για την καταπολέμηση της παράνομης μεύσης. Ε, πρέπει να θυμηθείτε ότι εμείς παρέχουμε μόνο στοιχεία όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Εκεί ε, κινούμεθα, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη μετανάστευση και για τη μεταναστευτική πολιτική. Στόχος μας είναι να είμαστε ο βασικός πάροχος πληροφοριών που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές, δηλαδή να δίνουμε την εικόνα των θαλασσίων μεταφορών. Όσον αφορά τα χωρικά ύδατα και τα σύνορα μεταξύ χωρών μένουμε εκτός αυτού. Από τη στιγμή που είναι ύδατα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εμείς έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε, αλλά δεν ανακατευόμαστε στο κατά πόσο τα ύδατα ανήκουν στο κράτος μέλος Α ή στο κράτος μέλος Β. Ευχαριστώ κύριε Ντιρόιτε. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, ο κύριος Ντερόιτε ε, θα μπορέσει να σας απαντήσει γραπτός. Στείλτε του ε, το ερώτημά σας στην ΕΜΣΑ είναι πολύ, ήταν πολύ συνεργάσιμος ε, όταν ήρθα σε επαφή εγώ μαζί του. Αλλά μας πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και που εξηγήσατε το ρόλο της ΕΜΣΑ στην Επιτροπή μας. Σας ευχόμαστε καλή τύχη για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας λέει ο κ. Διευθυντή. Θα έχει την υποστήριξή μα, λέει ο Πρόεδρο. Αναγνωρίζει ο κόσμο τη δουλειά που κάνετε. Και είναι καλύτερο να είμαστε δραστήριοι παρά να περιμένουμε να βυθιστεί κάποιο πλοίο για να δραστηριοποιηθούμε. Συγγνώμη. Αυτέ ήταν οι επικρίσει που ακουγόταν κατά το παρελθόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχουμε διορθώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πρόσκληση να επισκεφθούμε την ΕΜΣΑ. Σκεφτείτε το λοιπόν για να κανονίσουμε κάποια μελλοντική ημερομηνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα, διάλειμμα δύο λεπτών για να αλλάξουμε την διαρρύθμιση.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 Καθίστε παρακαλώ. Έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε σήμερα το πρωί τρία από τα τεν να συζητήσουμε. Πρώτο, ανταλλαγή απόψεων με το συντονιστή ΤΕΝ για το σχέδιο προτεραιότητας 3, τον κύριο Ταβινιό, που τον έχουμε μαζί μας σήμερα. The floor Κύριε Ταβινιό, έχετε το λόγο για κανένα δεκάλεπτο, άντε λίγο παραπάνω, αλλά αν ήσασταν δέκα λεπτά θα σας ήμασταν ευγνώμονες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μην σας φάω 4-10 λεπτά. Θα κάνω ό,τι μπορώ τέλος πάντων. Έχετε την έκθεση που έχω υποβάλει για την κατάσταση μετά από πέντε έτη εργασιών του τρίτου σχεδίου TEN που είναι όπως γνωρίζετε δύο διάδρομοι μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας και ένας διάδομος μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας. Όταν τελειώνει κανείς μια έκθεση μετά από πέντε χρόνια και έχει ιδιαίτερα το προνόμιο να περάσει την αρμοδιότητα ανανέωση του κύριο Σέκη, δεν στέκεται κανείς στις λεπτομέρειες. Περισσότερο κατα... στέκεται στα συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα αυτής της πενταετούς εργασίας ως υπεύθυνο μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων διαχειριστών και της Επιτροπής. Πρώτο συμπέρασμα πολύ θετικό είναι ότι η ανάγκη του σχεδίου προτεραιότητας αυτού γίνεται σήμερα ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Για έναν πολύ απλό λόγο. μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας οι δυσκολίες διέλευσης αυξάνονται και συσσωρεύονται, κάτι λογικό διότι υπάρχει μια χρονική προοπτική. Και δεύτερον, οι περιβαλλοντικές, ε, η περιβαλλοντική μέρημνα, οι περιβαλλοντικές διαστάσεις έχουν μεγαλύτερο μεγαλύτερη σημασία σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Είναι προφανές ότι οι συνδέσεις είναι ανεπαρκή και για τους επιβάτες ακόμα δεν περισσότερο για τα εμπορεύματα. Διότι κατά τη διάρκεια τη περίοδου αυτής εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν λιμένες που χρειάζονται ενδοχώρα. Άρα η σιδηροδρομική σύνδεση σήμερα είναι σημαντικότερη από ό,τι πριν. Δεύτερο συμπέρασμα, και δεν εκπλήσει, καθυστερήσαμε. Σε όλα τα μεγάλα έργα υπάρχουν καθυστερήσεις. Η διαπίστωση αυτή λοιπόν δεν πρέπει να μα οδηγείται και καλά σε απεσιοδοξία. Πρέπει να καταλάβουμε ωστόσο τους λόγους της καθυστέρησης. Οι λόγοι είναι, τουλάχιστον όπως τους εξέφρασα στην έκθεσή μου, συνθετικά τρει. Ένα. Ένα τεχνικό πρόβλημα. Για να κατασκευαστεί γραμμή υψηλής ταχύτητας χρειάζεται να κάνουμε σύραγγες, να περάσουμε δίπλα από πόλεις, να δημιουργηθούν υποδομές και να πάρουμε μια σειρά επιπλέον αδειών. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει πάντα μια σειρά κανόνων που πρέπει να τηρηθούν. Υπάρχουν διαβουλεύσεις που χρειάζεται να γίνουν. Οι διοικητικέ δομές δεν είναι ίδιες και από τις δύο πλευρές, αλλά παντού καθυστερούν. Δεύτερο θέμα, κάτι πολύ, δεύτερη αιτία, πολύ σημαντική για τα επόμενα έτη. Πρέπει να συνδυάσουμε τις εθνικές προτεραιότητες με τις διασυνοριακές προτεραιότητες. Και μόνο που το λέω νομίζω ότι καταλαβαίνετε τις δυσκολίες. Κάθε κυβέρνηση προφανώς ενδιαφέρεται περισσότερο για τη βελτίωση της εθνικής της υποδομής παρά για τις συνέπειες της βελτίωσης αυτής σε διασυνοριακές δομές. Άρα η σύσταση που περιλαμβάνει η έκθεση αυτή αναφέρει σαφώς ότι αν δεν μπορούμε να συνδυάσουμε τις εθνικές προτεραιότητες με την ευρωπαϊκή θα παραμείνει το πρόβλημα διότι η δημιουργία τέλεια μιας διασυνοριακής υποδομής με τη συνδρομή της Ένωσης για να διαπιστώσει κανείς μετά ότι το πρόβλημα πέρασε από το διασυνοριακό στο εθνικό δεν λύνουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι ο δεύτερος λόγος. Και αυτό με οδηγεί στο να κάνουμε, στο να κάνουμε μια σειρά προτάσεων, ώστε οι δομές στις οποίες μετέχουν οι Ισπανοί και Γάλλοι και ενδιαφερόμενες πλευρές, οι Ισπανοί και Πορτογάλοι και ενδιαφερόμενες πλευρές, θα πρέπει να εξετάζει όχι μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά όλη την υποδομή. Αν θέλουμε να φέρουμε κοντά τις προτεραιότητες, πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα εθνικά προβλήματα και τις διασυνοριακές διαστάσεις τους. Ζητάω λοιπόν από τις κυβερνήσεις να υπάρχουν ε, να υπάρξει μια νέα δομή στην οποία θα μετέχουν και οι συντονιστές και θα μπορούν να εξετάσουν κατά πόσον ε, όντως χρησιμοποιείται σωστά ε, ο προπολογισμό της Ένωσης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Η τρίτη δυσκολία αναφέρεται στην ανάγκη να εξετάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα υφιστάμενα δίκτυα πριν ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο δίκτυο. Αυτό είναι λογικό. Εντάξει, καθυστέρηση υπάρχει. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως με το υφιστάμενο δίκτυο. Πώς μπορούμε να καλύψουμε κάποιες από τις υφιστάμενες ανάγκες με το υφιστάμενο δίκτυο. Και ξέρετε εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και με τις εθνικές αρχές. Οι εθνικές αρχές θεωρούν ότι η δική μας αρμοδιότητα είναι μόνο το νέο σχέδιο και όχι ε, τα υφιστάμενα δίκτυα. Και εδώ προτείνουμε να μπορούμε να συζητούμε το σύνολο του ζητήμα, το, σύνολο των ζητημάτων μέσα στην δομή που προτείνω να δημιουργηθεί. Βεβαίως, ένα τέταρτο ημισημείο είναι το εξής. Ο κύριος Βίν, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος ε, για την σήμανση, θα έπρεπε να μπορεί να συμμετάσχει στις συζητήσεις αυτές, γιατί πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι συστάσεις γενικού χαρακτήρα για την διαλειτουργικότητα θα λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις αυτές και αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με τη συνεργασία του κ. Βίν, αλλά πρέπει να τον καλέσουμε. Και δύο ακόμα παρατηρήσεις, Πρόεδρε. Πρώτον, Στην υφιστάμενη κατάσταση που έχει τώρα, οι εργασίε στο ανάντι της διασυνοριακής δομής έχουν προχωρήσει περισσότερο στην Ισπανία από ό,τι στη Γαλλία. Παρόμοια είναι και η κατάσταση μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας. Παρότι η οικονομική κρίση γεννά κάποιες αβεβαιότητες για τα εθνικά προγράμματα σε ό,τι αφορά την δική τους ε, πλευρά του διαδρόμου. Δεύτερο σημαντικό σημείο όταν βλέπουμε όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ένωση βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση στη Γαλλία είναι περισσότερη από τη χρηματοδότηση στην Ισπανία και από την άλλη μεριά η χρηματοδότηση στην Ισπανία είναι περισσότερη από την χρηματοδότηση στην Πορτογαλία. Συμπερασματικά, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο σχέδιο. Δεύτερον, για να δώσουμε προτεραιότητα πρέπει να υπάρξει σημαντική πρόοδος τον επόμενο χρόνο το επόμενο, στο επόμενο χρονικό διάστημα και πρέπει να αλλάξει η δομή η σύνθεση των δομών συντονισμού μεταξύ Ισπανογάλων και, Γαλλο... και Ισπανοπορτογάλων. Από ό,τι ξέρω η Επιτροπή στο ξεκίνημα του νέου έτους θα κάνει τη νέα της πρόταση για τα διάφορα έργα προτεραιότητας και είναι προφανές ότι το οικονομικό πρόβλημα είναι κλειδί στην επιτυχία των έργων και δεύτερον η χρηματοδότηση πρέπει να πηγαίνει σε εκείνα τα έργα που έχουν προχωρήσει περισσότερο. Είναι πολύ δύσκολο το έργο, το ξέρει ο κύριος Σέκη, ε, θα το αντιμετωπίσει με χιούμορ και με ταλέντο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε για, μία, για ακόμα μία και τελευταία φορά. Να ευχηθώ στον κύριο Σέκη καλή επιτυχία στην υλοποίηση του, του ερώτητου αυτού έργου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Νταβινιόν. Πραγματικά ε, ανυπομονούμε για την καλή διάθεση και την εμπειρογνωμοσύνη του κυρίου Σακή. Ο κ. Γκράντε Πασκουάλ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Νταβινιόν. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνετε και πραγματικά το έργο που κάνατε το κληροδοτείτε στον κύριο Σάτσι και νομίζω ότι πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτό που κάνετε. Το καταλαβαίνουμε εμεί στο Κοινοβούλιο, διότι ξέρουμε ότι το κάνατε με εντιμότητα, αποτελεσματικότητα και σωστό τρόπο. Κρίμα που φεύγετε και κρίμα κυρίω που η δουλειά σα ε, συγκρούστηκε με κάποιου κάποιους αστάθμιτους παράγοντες που δεν είναι δική σας ευθύνη. Το λέω με ευγένεια αλλά με σαφή τρόπο για να μην υπάρχει σύγχυση. Είναι ασυγχώρητο να καταγγέλει στο μέλλον ο κύριος Σάτσι με τον ίδιο τρόπο, διπλωματικό τρόπο όπως και εσείς, την ανάγκη να είναι συμβιβάσιμο το έργο αυτό με το ευρωπαϊκό όραμα για να υπάρχει μια εσωτερική ε, να υπάρχει μια συμβατότητα μεταξύ του έργου και των εθνικών προτεραιοτήτων. Το σχέδιο 3 έχει τρία ε, διασυνοριακά βασικά στοιχεία την πορτογαλική διάσταση. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο έχει προχωρήσει, σίγουρα. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα προεκλογικού χαρακτήρα στη συζήτηση στην Πορτογαλία. Τα πορτογαλικά κόμματα θεμητά ε, ε, έφεσαν το ερωτηματικό του αν έπρεπε να υπάρχει μια εθνική προτεραιότητα ή όχι. Τέλο πάντων το, το ζήτημα λύθηκε και η Πορτογαλία δεν θα εγκαταλείψει το σχέδιο. Από την άλλη πλευρά, κάτι πολύ αρνητικό, είναι στο κομμάτι Γαλλία-Ισπανία. Το λέμε εξ αρχής. Έχουμε ένα χρέο στην Ισπανία, το λέω σαφώ. Μα βοηθάει στην αντιμετώπιση τη τρομοκρατία, είναι πολύ σημαντικό. Η αδελφική λοιπόν σχέση είναι δεδομένη. Δεν ισχύει το ίδιο ωστόσο σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον που δείχνει η Ισπανία στο να μην τελειώνει η Ευρώπη στα Πυρηναία. Θα έπρεπε να δώσει η Γαλλία μεγαλύτερη πώς το πει ζέση σε ένα σχέδιο που είναι ευρωπαϊκό. Η Ισπανία, το είπε ο κύριος ε, Νταβινιόν, τηρεί τις υποχρεώσεις, καταβάλει πόρου, πόρους πλήρως. Οι εργασίες ε, κλείνουν και νομίζω ότι αντιμετωπίζουν ωστόσο ένα κάποιο, ε, ε, μια κάποια έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς Γαλλίας που έχει άλλε άλλες προτεραιότητες. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Γιατί δεν είναι ένα ισπανικό έργο αυτό, αλλά ένα ευρωπαϊκό ουσιαστικό έργο ε, στη χώρα μας. Είναι καθοριστική σημασία. στο ίδιο και την Πορτογαλία. Άλλη αδελφή χώρα. Τα πυρηναία πρέπει να μπορούμε να τα περάσουν εύκολα γρήγορα και σωστά και επιβάτες και εμπορεύματα. Η καθυστέρηση σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εξάγουμε ό,τι μπορούμε να εξάγουμε και δεν μπορούμε να εισάγουμε ό,τι μπορούμε να εισάγουμε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί θέσατε το ζήτημα με σαφή τρόπο, χωρίς να κατηγορήσετε κανένα, ούτε κι εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βασικό ζήτημα είναι ότι το έργο αυτό έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Η δουλειά από πλευρά Γαλλία, η Ισπανία, συγγνώμη, έχει γίνει. Πιστεύω και η Γαλλία πρέπει να τηρήσει τι ε, υποχρεώσει τη λίγο λιγότερο στο Ερελαντή που θα είναι θετικό και για την Ευρώπη και για τις χώρες μας. Ευχαριστώ. Ο κ. Αλκαντράη για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νταβινιόν, καταρχάς σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την εργασία που κάνατε τα τελευταία πέντε χρόνια. Πρώτα μία γενική ερώτηση. Αναφερθήκατε σε κάποιες δυσκολίες και τονίσατε ότι πάνω από όλα ο καλύτερος συντονισμός είναι το κλειδί για την πραγματική πρόοδο. Μετά από πέντε χρόνια εμπειρίας μπορείτε να μας πείτε αν ως συντονιστής έχετε την αίσθηση ότι δεν έχετε αρκετά μέσα πίεσης των ανθρώπων, των διαφόρων εμπλεκόμενων ώστε να συνεργαστούν και να, να γίνει πρόοδος. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν μέσα χρηματοδοτικά και άλλα μέσα προπολογισμού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο ώστε η πρόοδος να είναι μεγαλύτερη και γρηγορότερη. Πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα. Μιλήσατε και για διαφορές μισολογικές και τα λοιπά. Η κυρία Μπιλμπάου για του άλλους. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Νταβινιό για τη δουλειά που έκανε. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό το έργο προτεραιότητας υπαριθμών 3 γιατί ζω σε μία περιοχή, τη χώρα των Βάσκων, όπου κατασκευάζεται το έργο και γνωρίζω συνεπώς τις δυσκολίες που είχαμε στο παρελθόν και τώρα. Για μας τουλάχιστον για τα βασικά θεσμι, για τα, τα θεσμικά όργανα της χώρας των Βάσκων, το έργο αυτό ήταν βασικό, γιατί απο, περιλαμβάνει τη σύνδεσή μας με την Ευρώπη. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε για να έρθουμε πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και ξέραμε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Σαρκοζή, ζήτησε να πραγματοποιηθεί μία έκθεση για να ξέρει, για να γνωρίζει κατά πόσον η αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ κάποιων δήμων, κάποιων οικολογικών οργανώσεων και κάποιων άλλων φορέων κατά της ε, σύνδεσης αυτής είναι, είναι, έχει βάση ή όχι. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για το τι θα γίνει, κατά, αν ε, η έκθεση που ζήτησε να του παρουσιαστεί ο Γάλλος πρόεδρος ε, είναι αρνητική για το κείμενο. Αν δηλαδή το συμπέρασμα είναι ότι η γραμμή που υπάρχει τώρα με κάποια, κάποιες βελτιώσεις θα ήταν αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες της Γαλλίας και αν αυτό θα συμπλήρωνε αυτό το ευρωπαϊκό έργο. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα χρειάζεται δεν, να γίνει κάτι, δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ε, φτάνει μια βελτίωση τη υφιστάμενη γραμμή. Θέλω να ξέρω ωστόσο ποια είναι η απόψή σα. Τι μπορούμε να κάνουμε εάν συμβεί αυτό το ενδεχόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Νταβινιόν για τις ε, προσπάθειές σας, ε, την υπομονή και τη διπλωματία σας. Όμως, Εξέτασα κάποιες από τις άλλες εκθέσεις που γράψατε τα προηγούμενα χρόνια και πραγματικά παντού αναφέρεται ότι είναι δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο και τώρα δίνεται ε, τα ενία στον διάδοχό σας. Ε, στην τελευταία έκθεση συγκεκριμένα αναφέρεται ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα αλλά δεν έχουμε επιτύχει τίποτα. Χτύπησαμε σε τείχο, δεν ε, πετύχαμε τίποτα. Και τώρα χρυσώνετε το χάπι, γιατί το κάνετε αυτό. Ο κύριος Κρέιμερ για τους πράσινους. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Την Παρασκευή είχαμε την έκθεση των συντονιστών και σήμερα πρέπει να συζητήσουμε. Εδώ τίθεται το θέμα πόσο χρόνο να να δώσω, ε, για να διαβάσω τις εκθέσεις όταν είναι στα αγγλικά και στα γαλλικά. Θα πρέπει λοιπόν για το μέλλον να έχουμε τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες για κάθε έκθεση και μετά να κάνουμε τη συζήτηση ώστε αυτοί που ενδιαφέρονται να μπορούν να διαβάσουν την έκθεση και να μην ε, περιορίζονται στην προφορική παρουσίαση. Αυτό για βάση. Δεύτερη παρατήρηση. Στην Γερμανία έχουμε και το Project 1, 2,5 εκατομμύρια, 15 χρόνια και πολύ μικρή επιτυχία. Ε, δεν ξέρω πραγματικά εάν ένα τέτοιο έργο που χρειάζεται 13 και 14 χρόνια για να γίνει, αν βοηθά και ειδικότερα με την αλλαγή του κλίματος ίσως με πιο σύντομα έργα να έχουμε επιτυχία. Στην Γαλλία και στην Ισπανία είπατε ότι υπάρχουν ε, προβλήματα. Αυτό έχει και προϊστορία. Υπήρχε μια εθνική οδός που πήγαινε μέχρι τα Πυρηναία και ταυτόχρονα ένας ε, σιδηροδρόμος ο οποίος όμως σταμάτησε. Εξαιτίας αυτού αποφασίσαμε τα χρήματα θα δίνονται μόνο όταν υπάρχουν διμερείς συμβάσεις ε, και δυνατότητα χρηματοδότησης ε, διμερείς. Μόνο τότε στέλνουμε χρήματα. Γι' αυτό ε, ρωτώ για τις δύο συνοριακές καταστάσεις στα Πυρηναία. Υπάρχει τέτοια διμερή σύμβαση μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή. Ε, η σύραγγα είναι πολύ επικίνδυνη εξαιτία της τρομοκρατίας. Είναι συγκεκριμένη γραμμή και πώς θα προχωρήσει και από τις δύο πλευρές. Τρίτο σημείο. Ε, η σιδηροδρομική σταθμή ΤΖΒ. Η Γαλλία έχει 10 και μόνο δύο ε, συνδέονται με γραμμές. Η Τουρ είναι μία περίπτωση. Είναι γρήγορα από την Τουρ μέχρι το Παρίσι, όμως ε, η άλλη πλευρά είναι πολύ αργή. Μόνο με το αυτοκίνητο μπορεί κανείς να πάει εκεί. Πώς γίνεται λοιπόν κανείς να θεωρεί ότι είναι σωστό αυτό να γίνεται όταν χάνει και χρόνο περνώντας μέσα από τις πόλεις. Αυτή ήταν η τελευταία μου ερώτηση. Έχω κι άλλες αλλά τις αφήνω. Ευχαριστώ. Το μόνο που θα πω εγώ, κύριε Νταβινιόν, είναι ότι αυτό το πρόβλημα δίνει την αίσθηση στα μέλη της Επιτροπής ότι το πρόβλημα είναι στη γαλλική πλευρά των συνόρων και όχι στην ισπανική. Και εσείς λίγο ακροθυγώς το αναφέρατε. Τώρα, αυτά τα προβλήματα είναι εθνικά. Προβλήματα είναι το πρόβλημα των σιδηροδρόμων ε, που πάντοτε σας δίνουν νέα λόγους που δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρά να σας δώσουν ένα λόγο γιατί μπορούν. Ότι πάντοτε δηλαδή δυσανασχετούν, ότι θεωρούν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα κτλ. Με αυτά κύριε Νταβινιόν ε, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω με την σειρά που τέθηκαν οι ερωτήσεις. Καταρχάς, Κύριε Ντεγκράντε Πασκουάλ. Εδώ και πέντε χρόνια είχαμε πρόβλημα με το γεγονός ότι δεν υπαρκούσε η κυκλοφορία πληροφοριών για την κατάσταση ως έχει, την πραγματικότητα. Επανέρχομαι στην ερώτηση του Προέδρου υπάρχουν και στοιχεία μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ανέφερε και αυτός. Και τα ομολόγο. Ε, ομολογώ. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα, όπως ξέρετε, ε, για πολύ καιρό διατηρήθηκε από την ισπανική πλευρά. Εμείς είχαμε κάποια ερωτήματα αν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα ή το άλλο ή αν θα καθυστερήσουμε. Όμως έλεγαν ότι θα τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα. Και πριν από δύο χρόνια μόλις, πολύ αργά καταφέραμε ότι θα ε, κατανοήσαμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει καθυστέρηση 5 έως 7 χρόνια. Έτσι λοιπόν ε, υπήρξε κάποια ένταση. Γιατί οι μεν εργάζονται επί μίας υποθέσεως ενώ ξέρουν ότι δεν θα τηρηθεί. Στην τελευταία μου λοιπόν έκθεση επέμεινα και είπα ότι αν δεν βελτιώσουμε την μόνιμη δομή συντονισμού πληροφορίας και διαφάνειας θα έχουμε ένα παλιό πρόβλημα όπως το πρόβλημα των συνδυοδρόμων να υποψιαζόμαστε το άλλο μέρος για προθέσεις που δεν θεωρούνται καλόβουλες τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν το έργο από τη μία πλευρά και από την άλλη εμποτίζεται με διάφορες τέτοιες ε, υποψίες. Όταν τελείωσα την ε, ε, πρακτική ανάλυση κατάλαβα τα εξής. Μεν, οι γαλλικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι το project αυτό είναι προτεραιότητα για αυτούς, παραμένει. Θα απαντήσω λοιπόν στην κυρία Μπιλμπάο ότι όντως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ένας Γάλλος υπουργός ανέφερε ότι υπήρχαν αμφιβολίες ε, για αυτή την προτεραιότητα ενώ ο Πρωθυπουργός διέψευσε. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε παραπάνω από αυτό. Εγώ ως άτομο, και αυτό απαντά στην ερώτηση που λέει γιατί δεν είπα ότι τα πράγματα είχαν τελειώσει, ότι εγώ ως άτομο έχω την αίσθηση ότι οι δύο πλευρές των συνόρων, όχι απαραίτητα για τους ίδιους λόγους, θέλουν ε, να έχουν ως προτεραιότητα να ρυθμίσουν τους λογαριασμούς τους. Ε, γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα τελειώσει αυτό το θέμα. Ναι, μεν υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θα ολοκληρωθεί το project. Υπάρχουν ή συγκεκριμένοι λόγοι που αφορούν τους Γάλλους και άλλοι συγκεκριμένοι λόγοι που αφορούν τους Ισπανούς ε, που θα τους κάνουν να επιτύχουν το αποτέλεσμα. Θα το πετύχουμε το αποτέλεσμα. Απλώς ε, πρέπει να βρούμε ποιες είναι οι λύσεις ε, και να μην μιλάμε στο κενό. Γιατί στο παρελθόν μιλούσαμε πολύ στο κενό, στον αέρα. Και γι' αυτό ε, έχουμε την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Όμως ε, δεν έχω αμφιβολίες, ούτε, καν, ούτε φόβους, ούτε καν για την Πορτογαλία. Βέβαια, η χρηματοδότηση σήμερα, δεδομένου των δημοσιονομικών προβλημάτων των κρατών, είναι ακόμα πιο δύσκολη από ό,τι στο παρελθόν. Όμως, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι ο ρόλος του συντονιστή είναι απλώς να μπορέσει να ρυθμίσει έτσι τα συμφέροντα και των δύο πλευρών ώστε να υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα. Αυτά είχα να πω για αυτό το θέμα. Για να απαντήσω στην κυρία Μπιλμπάου ή τέλος πάντων δεν θυμάμαι ποιος με έκανε την ερώτηση. Δεν υπάρχουν ε, διμερείς συμβάσεις μεταξύ Γαλλίας και Ισπανία. πέρα από αυτή που υπάρχει από το 1995. Δεν υπάρχει κάποιο καινούριο... Ε, και ο κύριος Κρέιμερ ρώτησε, ναι, ζητώ συγγνώμη. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο λοιπόν. Όμως, όπως λέω στην έκθεσή μου, θεωρώ ότι οι δομές διαχείρισης για αυτούς τους διαδρόμους δεν έχουν προσαρμοστεί Υπάρχει κάποια ομάδα αναφοράς, όμως ε, δεν έχουν ε, ρυθμιστεί και προσαρμοστεί οι απαιτήσει. Υπάρχουν συστάσεις φυσικά για αλλαγές που επί της αρχής έγιναν αποδεκτές από τις γαλλικές και ισπανικές αρχές. Θα δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστούν και αν. Φυσικά ο συντονιστής ε, θα είναι όντως ε, αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας, δεν θα τον προσκαλούμε απλώς ε, να έρχεται. Αυτό το διασφαλίσαμε τους τελευταίους μήνες και το διαπιστώσαμε. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα ψυχολογικό πρόβλημα, υπάρχουν αλληλοκατηγορίες που άλλες φορές ε, δεν έχουν βάση και άλλες όχι. Οπότε με τα στοιχεία που έχουμε πιστεύω ότι θα επιληθεί το πρόβλημα. Μια ερώτηση για το αν έχουμε αρκετή εξουσία εμείς ε, οι συντονιστές να κάνουμε τη δουλειά μας. Ο συντονιστής είναι ένας συντονιστής, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό δεν είναι εκπρόσωπος της Κομισιόν. Απλώς διευκολύνει. Και για να το κάνει φυσικά πρέπει να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Πλήρως. Αν ε, ε, διαβάσετε την έκθεσή μου θα καταλάβετε ότι αυτό δεν συνέβαινε τα τελευταία πέντε χρόνια. Όμως, με συμφωνία των δύο υπουργών με τους οποίους συναντήθηκα πριν γράψω την έκθεσή μου και μου δώσαν την άδεια να αλλάξω τη διαδικασία. Νομίζω ότι ο συντονιστής ε, πρέπει απλά να κάνει τη δουλειά του και να ε, αναφέρει στην έκθεσή του τι ακριβώς έκανε. Γι' αυτό οι αιτήσεις εκθέσεις είναι σημαντικές. Γιατί δείχνουν, δείχνουν τι έγινε, τι έπρεπε να γίνει και γιατί δεν συνέβη αυτό που έπρεπε να γίνει. Είναι λοιπόν ύψης της σημασίας για την Κομισιόν και το Συμβούλιο όταν αυτοί ε, θεσπίζουν τη δική τους θέση να συμπεριλαμβάνουν όλα αυτά τα στοιχεία γιατί η θέση της Κομισιόν σχετικά με τη Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία είναι αυτή που θα καθορίσει και την πολιτική τους. Και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει με βάση τις διάφορες προτάσεις των συντονιστών, του συντονιστών. Είπατε ότι και η διπλωματία και η υπομονή είναι καλή. Γιατί ε, δεν λέτε απλώς, ε, όμως μου λέτε, δεν μπορούν, δεν θέλουν κτλ. Δεν το έκανα γιατί δεν συμφωνώ. Μετά από πέντε χρόνια η εντύπωσή μου τελικά είναι ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να γίνει αυτό το project, μπορεί να γίνει, απλώς πρέπει να αλλάξουν οι μέθοδοι. Έκανα λοιπόν μία έκθεση η οποία μπορεί να χαρακτηρίζεται ως αισιόδοξη, όμως αυτό που λέει στην ουσία είναι ότι μπορεί να γίνουν περισσότερα από αυτά που έχουν γίνει. Και δεν είναι αδύνατο να γίνουν όλα αυτά. Ε, θα το έλεγα μόνο αν ήμουν πεπισμένος ότι είναι αδύνατο να γίνουν. Ε, δεν ξέρω, δεν είμαι πεπισμένο για κάτι τέτοιο. Ίσως ε, θα έπρεπε, δεν ξέρω, αλλά δεν είμαι. Μία από τις δυσκολίε κυρία Μπιλμπάου, είναι, είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί συνομιλητές. Αυτό το στοιχείο λοιπόν της ε, διαφάνειας και της ε, πληροφόρησης ισχύει και για τους ε, διάφορους ε, εκπροσώπους των χωρών αλλά και εντός των διαφόρων χωρών για όλους λοιπόν τους συνομιλητές. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι παρόντα στις συναντήσεις όπου κάνουμε το σχεδιασμό, θέτουμε τους στόχους και το κάνουμε τους ελέγχους. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να τους ελέγχουμε για να μπορεί η ίδια η Επιτροπή να ελέγξει αν θα συνεχίσει η ροή της χρηματοδότησης ή όχι. Είναι η Επιτροπή που λαμβάνει αυτή την απόφαση και ο συντονιστής είναι αυτός που πρέπει να πει αν είναι προτεραιότητα στο έργο, αν μπορούμε να υπερβούμε τις δυσκολίες, αλλά η πολιτική απόφαση είναι στα, στα χέρια των ε, πολιτικών αρχών, όχι στα χέρια του συντονιστή για τη διαθεσιμότητα της έκθεσης ε, στα χέρια των βουλευτών. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνο να απαντήσω. Εγώ εγκαίρως τελείωσα την έκθεσή μου. Μια τελευταία λέξη κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις δυσκολίες, τις αντικειμενικές δυσκολίες. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν ε, θέσαμε το... Όταν θέτουμε το χρονοδιάγραμμα, ε, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι υπεύθυνοι των σιδηροδρόμων είναι αυτοί που έχουν τις μηχανές, έχουν τα βαγόνια. Πρέπει επίσης να διασφαλίζουμε ότι υπάρχει λογιστική υποστήριξη και οι υποδομές και οι διαχειριστές ε, των τριών επιπέδων είναι διαφορετικοί. Ξέρετε ότι επειδή είναι χωριστέ αυτές οι αρχές, ο καθένα έχει τα δικά του προβλήματα και δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των άλλων. Ε, αυτό ισχύει και αλλού, αλλά πόσο μάλλον στους σιδηροδρόμους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Νταβινιόν. Και εδώ τελειώνουμε σας και πάμε στον κύριο Μπρίνκχορστ. Οπότε θα αλλάξουμε ξανά εδώ τους παρισταμένους στο Προεδρείο. Σας ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε και προσβλέπουμε σε μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω στο Προεδρείο τον κύριο Μπρίνκορστ. Έχει συνηθίσει να κάθεται σε τέτοια έδρανα. Έχει μεγάλη εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα 6 άξονας Λιούν Βουδαπέστης, Ουκρανία, μέχρι τα Ουκρανικά σύνορα. Κύριε Μπρίνκχορστ, έχετε 10 λεπτά. Uh, uh, Χαίρομαι που ξανάρθα στην Επιτροπή Μεταφορών. Ήταν σημαντικό σύμμαχος όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση και το όλο πρόγραμμα αυτό ωφελήθηκε από την ευρωπαϊκή προσέγγιση και ευχαριστώ που μου δίνει τη δυνατότητα να ξαναμιλήσω. Το πρόγραμμα αυτό το 6 είναι δύσκολο. Έχει μακρά ιστορία πολιτικών ζυμώσεων σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το 1994 συμφωνήσαμε στα πρώτα προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρχαν πολλά κοινά προβλήματα διασυνοριακής φύσεως που πλήττουν και τούτο. Δεν θα μακρηγορήσω. Θα, θα σας πω Ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί. Το Λιόν του Ρήνο. Το Ρήνο. δύο σημαντικές πόλεις από την γαλλική και ιταλική πλευρά. συνδεόταν επί σειρά ετών, αλλά υπάρχουν και φυσικά φράγματα. Από την ε, γαλλική πλευρά υπάρχει πρόοδος θετικές εξελίξεις στη Γαλλία. Έγιναν τρεις διερευνητικές σύραγγες. Θα είναι έτοιμες στο τέλος του χρόνου. Σε Μαρτέν Λαπόρτ είναι η πρώτη σύραγγα. Λαπράζ και μετά το Μαντάν. Στην Ιταλία, όπως θα θυμόσαστε, το παρατηρητήριο εκεί ε, βρήκε λύση για την ευθυγράμμιση. Πρέπει να αναμειχθούν κάποιοι δήμοι. Είχαμε πολλά προβλήματα, βλέπετε, στην Βαλέ de Suze. Και τελικά δεν φτιάξαμε το κομμάτι του σιδηροδρομικού που θέλαμε εκεί. Ελπίζω οι Ιταλοί να λύσουν το πρόβλημα μέχρι το Δεκέμβριο. Και οι ερευνητικέ εργασίε από πλευρά Ιταλία να ξεκινήσουν αρχέ του επομένου έτου. Και να προσημειωθούν και τα σχετικά κονδύλια. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των κονδυλίων. Αυτή είναι η μακροπρόθεσμο όραμα για τη νέα σύραγγα μεταξύ Λιών και Τωρίνου. Θα είναι 57 χιλιόμετρα μήκος, είναι μεγαλύτερη σύραγγα ακόμα και πιο μακριά σύνταγα από, την διόρυγα, από τη σύραγγα που ενώνει ε, Βρετανία με Γαλλία. Τα μέλη λοιπόν στις διακοπές κάντε ένα ταξιδάκι από Λιόν στο Τωρίνο να δείτε είναι πολύ ωραίο το τοπίο αλλά χρειάζεται πολλές ώρες η παρούσα γραμμή και περί αυτού πρόκειται. Αν η παρούσα ε, γραμμή δεν κερδίσει μερίδιο στην κυκλοφορία θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τη νέα γραμμή να είναι βιώσιμη οικονομικά για να μπορέσουν να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους οι επενδυτές. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία. Για να λειτουργήσει αυτή η διασύνδεση διαμέσου των άλπων μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. Για τη λύση του προβλήματος δημιουργήθηκε μια ομάδα υψηλού επίπεδου όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και οι ρυθμιστικές αρχές συμμετέχουν ακόμα. Να πω και το εξή. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδεοδρόμων που δημιουργήθηκε προετών ε, πρέπει να δούμε ότι δραματίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Λειτουργεί για το ERTMS επίσης. Αλλά εδώ έχουμε πιλωτικό πρόγραμμα που συνεργάζονται όλοι οι φορείς στενά. Υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη. Και γι' αυτό ελπίζω θα πετύχουμε καλύτερη διαλειτουργικότητα και συντονισμό μεταξύ των δύο εθνικών δικτύων. Πρόεδρε, σε πρώτερες συζητήσεις θέλαμε να εντοπίσουμε τις δυσκολίες. Δεν θα σας κρυφτώ. Έχω λειτουργήσει σε πολλούς, έχω κινηθεί σε πολλούς ζωή μου Στου σιδηροδρόμους όμω, η εσωτερική αγορά δεν έχει διεισδύσει. Κυρίως αυτού που παίρνουν τι αποφάσεις. Από Χάγη ήρθα Βρυξέλλε σήμερα. Το κάνω πάντα αυτό. Και πάλι καθυστέρη 40 λεπτά είχα. Διότι δεν έχει προτεραιότητα το νόμο. Τους αρέσει καλή διασύνδεση Ανατολή με Δύση και αυτή η διασύνδεση δεν έχει τόσο μεγάλη προτεραιότητα. Θέλει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδεδρόμων να συμμετάσχει. Ξέρει πολλά, έχει μεγάλη εμπειρία Λοιπόν, σημαντική είναι η διαλειτουργικότητα. Έχουμε αναφερθεί σε αυτού. Και επίσης αλλαγή από ράγε μεταξύ στα σύνορα. Υπάρχει λοιπόν διαφορά στις ράγες και γι' αυτό δεν περνάνε τα τρένα εύκολα. και θα πρέπει οι ατομομηχανέ ε, να μπορούν να κινούνται και δύο πλευρέ των σύνορων. Επίση, η σηματοδότηση διαφέρει μεταξύ Γαλλία και Ιταλία. Και η επικοινωνία είναι πολύ δύσκολη. Και πρέπει να αλλάξει ο μηχανοδηγό στα σύνορα. Όχι μόνο η μηχανή. Και αυτό χρειάζεται χρόνο. Και πρέπει να δοθούν με τα χέρια από τον ένα στον άλλο διάφορα έγγραφα όταν παραδίδεται η ατμομηχανή. Όπως σας είπα δεν είχα ανακατευθεί με τους ιοδρόμους κατά παρελθόν και σαν συντονιστής μου αρέσει να βλέπω πώς λειτουργεί στην πράξη Ευρώπη. Αυτά είναι τα ζητήματα. Και εδώ μπορεί να κάνετε διαφορά στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το ιστορικό. Χρειάζεται συγκεκριμένη δουλειά. Δεν έχω παράπονα. Και στη Γαλλία και στην Ιταλία αρχίζουν να καταλαβαίνουν τα διακυβευόμενα. Ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Η Ευρώπη αν δεν αλλάξουμε τα, την κατάσταση δεν θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, το Ρήνο ταιριέστη. Ενθαρρυντικά τα πράγματα. Υπάρχει έλλειψη πρόοδου στο κομμάτι μεταξύ Βενετίας και Τεργέστης. Και αν δεν δημιουργηθεί αυτή η γραμμή, δεν θα προχωρήσει το πρόγραμμα και δεν θα προσελκύσουμε και κονδύλια. Το PP6, το πρόγραμμα 6, δεν είναι μόνο κάτι που αφορά την Γαλλία και Ιταλία, αλλά Ανατολή με Δύση είναι η διασύνδεση κεντρικής Ευρώπης με δυτική Ευρώπη, νοτίως των Άλπαιων. Και πρέπει να γίνει η διασύνδεση τεριές της Βενετίας. Βλέπω κάποιος από τη Βενετία εδώ και ελπίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου. Τεργέστη και κόρποτε φράτσα. Γίνεται συνεργασία μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας για τη σύνδεση με τον Τιβάτσα, αλλά η πρόοδος έχει κολλήσει. Η Τεργέστη κάποτε ήταν κατεχόμενη και είναι στη γωνία της Ιταλίας και ξαφνικά από εκεί που ήταν κάπως απομονωμένη από την Ιταλία το αρχίζει να ξανασυνδέεται με την Ιταλία. Χρειάζεται βήμα συγκεκριμένο. Χρειάζονται κοινέ δομές όπως είχαμε για Λιόν, Τωρίνο και Σαμπερί και θα πρέπει στην Τεργέστη να υπάρξει κοινή υποδομή Σλοβενίας-Ιταλίας. Χρειάζομαι βοήθεια. Το παρελθόν πρέπει να μείνει στο παρελθόν. Να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Και μετά έχουμε το Τιβάτσα, Λουμπριάνα, Βουδαπέστη. Πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Κάντε το ταξιδάκι, πάρτε το τρένο από την Τεργέστη, πηγαίνετε στη Βουδαπέστη και πάρτε μεγάλο βιβλίο πόλεμος Κυρίν του Τολστόη, πάει κουτί, ας έρθει κουτί. Μέχρι θα στη Βουδαπέστη θα το έχετε ξεπετάξει. Και εγώ θα σας βοηθήσω για να το κάνετε αυτό πιο θετικέ εξελίξει σήμερα όμω, διότι οι Ουγγαροί και οι Σλοβαίνοι καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται να συνεργαστούν. Αλλά έχουν πληγεί από την κρίση τα κράτη-μέλη, βλέπετε. Και για πρώτη φορά οι Σλοβαίνοι και οι Ούγγροι κάνουν πρώτα βήματα για την υλοποίηση του κοινού προγράμματο. Ποια είναι η γενική μου αξιολόγηση. Ενθαρρυντική πρόοδο έχει επιτευχθεί, παρόλο που περνάμε δύσκολου οικονομικού καιρού. Χαλεπού. Βεργαίνει, ταιριέστη, ε, Ταιριέ κόπερ κόπε με ανησυχεί, σαν να πηγαίνει μουλάρι είναι. Και το ταιριέ Βενετία με ανησυχεί. Πέντε χιλιόμετρα. βλέπεις την Τεργέστη, κόπερ Τεργέστη. Δεν υπάρχει δρόμος όμως κανονικά. Άντε να καταλάβουν ότι χρειάζεται διά, ε, σιδηρόδρομος. Και θέματα οικονομικά τίθενται τα οικονομικά θέματα. Οικονομική κρίση περνάμε, το ξέρουμε. Οι υποδομές χρειάζονται, εξυπηρετούν την Ευρώπη. Αλλά τα κράτη-μέλη έχουν μείνει άφραγκα. Δημόσια επενδύσεις δεν έρχονται. Αλλά επανέρχεται η κοινή λογική μετά από ένα χρόνο κρίσης. Οι επενδυτέ βλέπουν ότι μπορούν να έχουν κέρδη μακροπρόθεσμα. Θα αναλάβω μια πρωτοβουλία έναντι τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χρειάζομαι τη βοήθειά σα. Θα ήθελα ένα σχέδιο στο οποίο συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να υλοποιηθούν οι παρέτες υποδομές που είναι δαπανηρές. η ενέργεια και οι υποδομέ είναι κάτι σημαντικό. Και γιατί έχουμε μείνει πίσω όσον αφορά τι υποδομέ των σιδηροδρόμων. Όχι δεν ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά χρειάζεται εσεί να πιέσετε περισσότερο τα κράτη-μέλη. Για να αλλάξουν οι εθνικέ συνήθειε και νοοτροπία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να ελκύσει και άλλου επενδύτε. Και έτσι μπορεί να υλοποιηθούν τα προγράμματα. Χρειάζεται εστιασμένη χρηματοδότηση. Να λειτουργεί εσωτερική αγορά με υπεύθυνο περιβαλλοντικά τρόπο. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εμπλακή, Μελλοντικέ δραστηριότητε. Δεν φεύγω από τη δουλειά. Ανανεώθηκε η θητεία μου μέχρι το 2013. Πρέπει να με ανεχθείτε, φοβάμαι. Χρειάζονται λοιπόν χρήματα. Πρώτο στόχο για κάποια κομμάτια. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων. Θέλω να κινητοποιήσω, να ενδιαφερθείτε. Πάτε το τρένο Λιόν Τωρίνο, είναι ωραία διαδρομή. Αλλά θα καταλάβετε τότε γιατί είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε αποτελέσματα. Δεν παρετούμεθα. Αλλάζουμε σταδιακά τα πράγματα. Αλλά όπω όλα, στην Ευρώπη προχωρούν αργά τα πράγματα. Χρειάστηκε 10 χρόνια η συνθήκη τη Αβώνα. 15 χρόνια θα χρειαστεί το τρένο. Και μέχρι τότε ελπίζω να είμαι ακόμα ζωντανό. Ευχαριστώ κύριε Μπρίνκχορστ. Πριν δώσω το λόγο στους αγορητές που έχουν ζητήσει το λόγο, εγώ επί σειρά ετών ήμουν ανακατεμένος στους σιδηροδρόμους και θέλω να πω ότι και εγώ είχα απογοητευτεί όσο και εσείς για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα τρένα. Εσείς διασκεδάζετε, εγώ όμως απογοητεύομαι και θυμώνω. Αργός, πολύ αργός ο ρυθμός με τον οποίο κινούνται στη σιδηροδρομοί. Να πω και μια, μια ιστορία ανεκδοτικά. Πολλοί βουλευτές ξέρουν ότι αγαπώ τους ιδοδρόμους. Υπάρχει ατμομηχανή. Το Flying Scotsman, ο υπτάμενος Σκοτσέζος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και θέλαν να ξαναφτιάξουν τον υπτάμενο Σκοτσέζο, την ατμομηχανή. Τον έκαναν όλοι, είπαν φανταστικό πρόγραμμα. Και όλοι οι σιδηρόδρομοι μπλέξανε κατά πόσο είχαν βάψει σωστό χρώμα, τη σωστή απόχρωση του πράσινου την ατομηχανή. Αυτή, αυτή τη φρούστρα νιώθουμε όταν εργαζόμαστε σε αυτό το τομέα στους σιδηροδρόμους. Αλλά κύριε Μπρίγχορστ, μπορώ και εγώ να βοηθήσω να πιέσουμε για να πετύχουμε το θαύμα ανοιχτή αγοράς, εσωτερικής αγοράς των σιδηροδρόμων. Και πιστέψτε με, χρειάζεται αποφασιστικό αλλά πιστεύω ότι κάποια μέρα θα υλοποιηθεί ο στόχος. Τώρα αν θα ζω, όταν συμβεί αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Θα συμβεί όμω κάποτε. Εντάξει, έχουμε τέσσερι αγορητές. Ελκ, κύριο Κάντσιν, ο πρώτο. Πόσο χρόνο θα έχω, Πρόεδρε, εκτός μικροφώνου Πρόεδρος. <laughs> Αν αυτό ήταν το πρώτο, να σας πω διακόπτει ο πρόεδρος. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται και η κυρία Λίχτεμπεργκ, η οποία έχει έναν, ε, ένα βιβλίο με δρομολόγια τρένων. Προσοχή. Έλεγα λοιπόν ότι ξεκινήσαμε το 1994 να μιλάμε για το έργο αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να το προσέξουμε κάπως περισσότερο. Η κατάσταση είναι θλιβερή. Και για την υποδομή αυτή καθεαυτή, αλλά και για την οικονομία που χρειαζόμαστε σχετικά, γιατί η κατάσταση δεν είναι και ιδιαίτερα θετική στον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που θα μπορούσαμε και να λύσουμε ωστόσο. Εγώ κάνω μια γενική συζήτηση, μια γενική παρατήρηση και μετά θα μπω στα επιμέρους. Θίξετε μια σειρά σημείων. Το πρόβλημα είναι χάραξης, πρόβλημα χάραξης, πρόβλημα πολιτικών επιλογών. Εγώ ξέρετε είμαι από τη Βενετία. Το ξέρω το ζήτημα από καιρό. ήταν το Τωρίνο Λιόν, ήταν το Βενετία Ντιβάτσα και το, η διαδρομή μέχρι τη, χάραξη μέχρι τη Λουμπλιάνα. Εάν είναι πρόβλημα χάραξης και πολιτικών επιλογών, πρέπει να είμαστε πολύ πιο κάθετοι και να έχουμε περισσότερες εξουσίες για να μην ε, δίνουμε στην τοπική αυτή περιφερειακή αυτοδιοίκηση επιλογές που δεν τις ανήκουν. Εμείς θα πρέπει να καταφέρουμε να κλείσουμε και να δώσουμε μια, ένα προγραμματικό ορισμό ξεκινώντας από εκεί και πέρα. Εγώ νομίζω ότι ένα σοβαρός προγραμματισμός περιλαμβάνει ροές και κόμβους. Μεταξύ των ροών και των κόμβων πρέπει να κατασκευάσουμε τον προγραμματισμό, να φτιάξουμε τον προγραμματισμό μας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που ήθελα να υπογραμμίσω. Το δεύτερο αφορά τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια εξαιρετική τεράστια ε, απέτηση. Ξεκινάμε από το 3 που συζητήσαμε προηγουμένως, τελειώνουμε στη Βουδαπέστη και το Κίεβο με, με, με έναν άλλο δρόμο, ενώ μας διασχίζουν κάθετα άλλοι μεγάλοι ο άξονα Βαλτικής, ε, Αδριατική, ο, ο, και ο 24. Τρει βασικοί, τρεις, βασικοί άξονες κάθετοι λοιπόν βορανότου. Οι διαδικασίε και ο χρόνος υλοποίησή του τους συνδέονται κατά βάση με την πολιτική μας βούληση. Το άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης το άφησα τελευταίο, αλλά πιστεύω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε οικονομικές λύσεις. Εγώ προτείνω κάτι που θα μπορούσε να είναι πέραν των ομολόγων που άκουσαν, για τα οποία άκουσαν να γίνεται λόγος και που μετά διασπαθίζονται από εδώ και από εκεί, θα ήθελα να υπογραμμίσω την πρόταση δημιουργίας ενός ταμείου ακριβώς για τις υποδομές αυτές. Ιδέες αυτή που τη θεωρώ σημαντική. Το Ταμείο αυτό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μετέχει σε project financing κα, κατά μήκο των ε, επιμέρους ε, διαδρόμων. Μόνα τους δεν επιβιώνουν τα σχέδια. Δεν συμπληρώνεται το business plan. Δεν υπάρχουν τοπικοί πόροι. Πιστεύω ότι μια πολιτική που διαμορφώνεται με τον τρόπο αυτό θα επέτρεπε να λειτουργήσει ένας μηχανισμός που θα επέτρεπε έναν, ε, μια χρηματοδότηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσω των ΣΔΙΤ για την χρηματοδότηση επιμέρους υποδομών και για να υπάρξει ένα ενιαίο και συμπαγές σύστημα χρηματοδότησης γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό τώρα να ξεκινήσουν οι, πρωτοβου... οι δημόσιες αυτές πρωτοβουλίες και να στηριχθούν βεβαίως από ιδιώτες. Άρα να πάρει μπρο και ο μηχανισμός ιδιωτικής χρηματοδότησης. Θα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που μιλήσαμε προηγουμένω. Τέλο πάντων, κλείνουμε ένα πολύ σημαντικό και ειδικό πέρασμα ώστε να ξεκινήσει το σύνολο. Θα σταματήσω γιατί με απειλεί με το σφυρί το πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές κύριε Τικάου. Τρία λεπτά Σίλβια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Σύντομη. Έχω μία ερώτηση. δεν αφορά μόνο το 6 αλλά και το 17 σχέδιο προτεραιότητας. Ελπίζω στο μέλλον τα δύο αυτά έργα να γίνουν, να ενωθούν κάπου γύρω από τη Βουδαπέστη και να επεκταθούν και προς το Βουκουρέστι και την Κωνσταντζα. Διότι μόνο έτσι θα υπάρξει η υποδομή τρένων υψηλής ταχύτητας που θα καλύπτει όλη την Ένωση. Η ερώτησή μου είναι, τι όραμα έχετε εσείς. Θα υποστηρίζετε αυτό το φιλόδοξο έργο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το 6 πρώτα στη Βουδαπέστη και μετά μέχρι το Βουκουρέστη και την Κωνσταντζα. Η κύριε Λίχτεμπεργκερ. Τρία λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για τους χάρτες. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι σε αυτό το project πρέπει να πούμε καταρχάς ότι είναι κάτι διαφορετικό να ε, συζητάμε για τους σιδηροδρόμους ε, της Ιταλίας και να τους χρησιμοποιούμε. Εγώ συχνά κάνω και τα δύο. Να μιλήσω αγγλικά. Τυρολέζικα. Δεν έχουμε διερμηνέα για τυρολέζικα. Θα συνεχίσω στα αγγλικά λοιπόν. Μπορείτε να συνεχίσετε στα γερμανικά. Ωραία. Δεν θέλω να μου το βγάλετε από το χρόνο μου. Άρα η χρήση των σιδηροδρόμων στην Ιταλία είναι ένα πρόβλημα πάντοτε και θα ήθελα λοιπόν να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα σε αυτή την περίπτωση. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποια κρίσιμα σημεία, λιών τορίνο, η Σύραγγα είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο και κρίσιμο. Αλλά έχουμε και ανατολικά, νοτιοανατολικά και βόρειο-ανατολικά της Βενετίας ένα κομμάτι. Όταν θέλουμε να κάνουμε γενικά ελκυστικούς τους σιδηροδρόμους δεν θα πρέπει να πάμε σαν υπνοτισμένοι και να κολλάμε μόνο σε αυτά τα δύο σημεία να κοιτάμε τουλάχιστον το ενδιάμεσο όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και στην πραγματικότητα να είναι αρκετά ελκυστικό για τους χρήστες. Αυτό για μένα είναι η βάση και γι' αυτό είναι σημαντικό να λέμε ότι όταν σκεφτόμαστε τους κοινούς ευρωπαϊκούς διαδρόμους θα πρέπει να σκεφτόμαστε τα κοινά σημεία, να μην κολλάμε σε μεγάλα project αλλά γενικά να κοιτάμε τα κομμάτια της υποδομής μεταξύ αυτών των κρίσιμων σημείων και να προσπαθούμε αυτά να τα κάνουμε προσβάσιμα και ελκυστικά. Τότε θα μπορέσουμε να έχουμε δικαιολογία, να κάνουμε τεράστια χρηματοδότηση, να δώσουμε χρήματα δηλαδή για αυτές τις μεγάλες σύραγγες. Όμως αν φτιάχνουμε μόνο αυτές τις σύραγγες, ε, όπως είπε στο παρελθόν και ο κύριος Κουστάτσα, ε, είναι σαν να χτίζεις την έρημο παλάτια. σε περίπτωση λοιπόν που οι γραμμές ε, που συνδέουν τους μεγάλους ε, κόμβους ε, δεν είναι απλώς εξαίρεση, δεν θα έχουμε, θα έχουμε... Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι λοιπόν μεγάλο θέμα. Να δούμε ποια είναι τα σημεία που μπορούμε ήδη να χρησιμοποιήσουμε και μετά να δούμε όλες τις περιστάσεις ε, που θα οδηγήσουν ε, στη διέλευση από τα κρίσιμα σημεία. Τώρα ε, έχουμε την εντύπωση στον κόσμο ότι φτιάχνουμε μια σύραγγα, δεξιά-αριστερά δεν υπάρχει τίποτα. Τι είναι αυτό το πράγμα τελικά. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε εμπλέξει τον κόσμο στην περιοχή. Θεωρούν ότι δεν αφορά αυτούς αυτό το θέμα θεωρούν ότι κάποιον άλλον ε, ε, Ολλανδό, ας πούμε, εξυπηρετούν, χωρίς να φύγω τους Ολλανδούς, που θέλει να πάει από την Άπολη στην Ολλανδία, ξέρω εγώ. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε μαζί μας ε, τους ντόπιου και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί δεν θεωρείται ότι έχει νόημα αυτό το project. Έτσι λοιπόν ε, αυτό συνέβη και περιπτώσεις που κάποιες ε, γραμμές ας πούμε κυρώθηκαν και προσπαθούμε τώρα να τις παρακάμψουμε. Αυτό είναι γενικά το πρόβλημα στην Ιταλία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαντάλεν. Από τους ιδιωτικούς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχετε μακρά εμπειρία ως επαγγελματίας κύριε Μπρινκότς φαντάζομαι ότι αυτό είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές που αναλάβατε. Σας θαυμάζω γιατί πραγματικά δείχνετε ότι απολαμβάνετε. Ξέρετε, το κράτος ήταν τόσο πολύ και για τόσο πολύ καιρό κυρίαρχο στους ιδεδρόμους που είναι δύσκολο να το δούμε ε, ως μια επιχείρηση όπως κάθε άλλη. Είπα λοιπόν ότι, έλεγα λοιπόν ότι δουλε, πραγματικά κάνετε μια από τις πιο δύσκολες δουλειές στις, στη ζωή σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Διάβασα την ε, προηγούμενη έκθεσή σας για το κομμάτι Copper Divacha που θα ξεκινούσε το 8. Τώρα βλέπω στη δική σας έκθεση ότι δεν ξεκίνησε αυτό το κομμάτι. Άρα μιλάμε για μεγάλες καθυστερήσεις. Γιατί δεν ξεκίνησε η δουλειά. Τον Τολστόι διαβάζουν οι υπεύθυνοι. Δεύτερον, εσείς ως συντονιστής είστε αισιόδοξο. Πιστεύετε ότι θα γίνει. Άντε, πήρε μπρο, αλλά νομίζετε ότι θα κλείσει, θα ολοκληρωθεί. Πιστεύετε ότι θα πετύχει αυτή η διοσυνοριακή σύνδεση. Δύο ακόμα ομιλητές υπάρχουν. Η κυρία Ντολτέ επανέρχομαι σε αυτά που είπαν κάποιοι προηγουμένω για την συμμετοχή του πληθυσμού και το ενδιαφέρον του πληθυσμού για το έργο αυτό. Στο κομμάτι Λιών Τωρίνο, ο πληθυσμό στη γαλλική πλευρά αναμένει με ανυπομονησία και πολιτικά υπάρχει απόλυτη ομοφωνία. Βεβαίως είχαμε και το προηγούμενο της του ατυχήματος στο τούνελ του Λευκόρου στο Οδικό και στο Φρεζής. Ξέρουμε ότι το πέρασμα των Άλπαιων έχει τεράστιες απαράδεκτες καθυστερήσεις, λιγότερο το 9 λόγω της κρίσης, αλλά το 7 στον αυτοκινητόδρομο υπάρχει, από τη Λιόν μέχρι τα τελικά σύνορα, υπάρχει ένα, ε, μια σειρά, ε, μια ουρά φωτιγών συνεχώς. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι πρέπει να περάσει στις Άλπεις τουλάχιστον όσο περισσότερο κυκλοφορία γίνεται από το δρόμο στο τρένο. Αυτό τεχνικά μπορεί να γίνει. Ο τύπος ε, τις τελευταίες ε, μέρες αναφέρεται, αναφέρθηκε στο ότι υπάρχει μια αντίθεση του πληθυσμού στην Ιταλική πλευρά. Τι άποψη έχετε. Τελευταίος ο κύριος Κράμερ εδώ ε, μάλλον έχει να κάνει όχι τόσο με χρήματα. Είπατε ότι χρειάζονται χρήματα. Πρέπει να πει πιο γρήγορα η έρευνα. Υπάρχει αυτό το κοινό, κενό 5 ε, χιλιόμετρων. Δεν είναι λοιπόν μόνο τα χρήματα, είναι και η καλή θέληση. Θα πρέπει καταρχάς λοιπόν να φτιάξουμε αυτό που είναι γρήγορα εύκολο να γίνει για να επικεντρωθούμε μετά στα κενά ε, και να έχουμε την υποστήριξη του κοινού. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη. Για τη σύνδεση με τη Βουδαπέστη υπάρχουν και άλλες ε, εναλλακτικές, ε, Παρίσι, Μπρατισράβα. Ο κύριος Μπάλαστη ήταν συντονιστής και ήθελε να συμπεριλάβει τη χώρα του. Αυτό ήταν χαζό. Και στην Βουδαπέστη και στη Βρατισλάβα όλοι το ίδιο σκέφτονται. Όμως επειδή είναι Ούγγρος, γι' αυτό έγινε. Υπάρχουν και σε άλλες περιπτώσεις ε, που έγινε αυτό. Είναι χαζή αυτή η διαδικασία όμως που ακολουθείται. Αυτό το θέμα της σύνδεση μέχρι τη Βουδαπέστη θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό όμως που μου λείπει εμένα είναι γιατί υπάρχει πρόβλημα μεταξύ ταιριές της ΚΟΠΑ γιατί υπάρχουν δυσκολίες, πού μπορούμε να βοηθήσουμε τέλος πάντων. Okay, thank you, Michael. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρίνκος, θα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ όλα τα μέλη για τις ερωτήσεις. Πάντα βοηθούν οι ερωτήσεις αυτές των συντονιστή. Καταρχάς, είναι σημαντικό να αναλύσουμε. Το είπε και η κυρία και Πρέπει να έχουμε μια εικόνα του συνόλου. Ο κ. Βαμπάλεν είπε ότι είχα μεγάλη καριέρα και να σας πω την αλήθεια, εάν δεν είχα μια εικόνα συνολική δεν θα αναλάμβανα τη δουλειά αυτή. Δεν, θα, δεν θέλω να ε, ασχοληθώ μόνο με το κομμάτι Λιών Τωρίνο, αλλά να ενώσω την Δυτική με την Αντουργή Ευρώπη. Είχα πάντα ένα όραμα. Ο κύριος Βαμπάλεν ανοίξει άλλο πολιτικό κόμμα, αλλά πρέπει να πιστεύουμε ότι αν θέλεις να πετύχεις το όραμά σου πρέπει να έχεις μια συνολική οπτική. Δίκιο έχετε όταν λέτε ότι το θέμα είναι εθνικό, τοπικό και περιφερειακό ταυτόχρονα, γιατί και η Ευρώπη έτσι είναι. Υπάρχουν ωστόσο σε όλες τις χώρες τοπικά θέματα Είτε μιλάμε για περιβάλλον, είτε μιλάμε για πυρηνικού σταθμού, παντού υπάρχει η τοπική διάσταση που λέει όχι, όχι, όχι στο, στο δίπλα μου, μακριά. Αν θέλετε λοιπόν να πετύχετε κάτι χρήσιμο, καλό θα ήταν να πάτε στην κοιλάδα Σούσα, να μιλήσετε με τον κόσμο εκεί. Δεν εγκαταλείφθηκε το πρόγραμμα από την καινούργια κυβέρνηση. Τώρα η υποστήριξη είναι μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά δεν έχουμε κλείσει την κατάσταση. Μέχρι τον Νοέμβριο, Νοέμβριο έχουν περιφερειακές εκλογές. Μέχρι να κλείσει, μέχρι να τελειώσουν και οι εκλογές, δεν είμαι σίγουρος ότι ε, θα κλείσει. Τώρα, με μου λέγατε να γίνει ένα νέο ταμείο. Θα σα απαντούσα όχι. Αλλά το τι μπορούμε να κάνουμε τώρα μπορώ να σα το πω. Να μιλήσουμε με την κυβέρνηση, μπα και τα βρούμε με τι τοπικέ αρχέ. Αυτή είναι η εικόνα μου. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Το πρόβλημα στο Λιόν Τωρίνο δεν είναι το τούνελ, αλλά η βελτίωση της τωρινής κατάστασης. Γι' αυτό και ο οργανισμός σιδηροδρόμων, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμός Σιδηροδρόμων είναι χρήσιμο. Υπάρχουν μια σειρά διαστάσεων που δεν τι είχα σκεφτεί ποτέ. Με ρωτήσετε, είμαι αισιόδοξο, είμαι. Και πιστεύω, διότι πιστεύω στο σχέδιο, διότι βασίστηκα στη βιωσιμότητα. Ήμουν Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντο 7 χρόνια. Κανεί δεν μιλά για το περιβάλλον τότε, κανεί δεν μιλούσε για το περιβάλλον, τότε παρά μόνο κάποιοι πράσινοι. Τώρα όλοι μιλάνε για το περιβάλλον. Ε, αλλά το πρόβλημα είναι ο εθνικισμός. Οι εθνικές συνοδομικές επιχειρήσεις το μόνο που πιστεύουν είναι ότι ο κόσμος τελειώνει στα σύνορά τους. Εσείς είστε οι μόνοι που βλέπετε το διευρωπαϊκό. Τώρα για τα συγκεκριμένα θέματα. Κύριε Καντσιάν, όντως υπάρχουν προβλήματα χάραξης και βοηθήστε με και στην Σούσα και στο κομμάτι Βενετία Τεργέστη. Ο κύριος Μορέτη είναι το αφεντικό των τρένων στην Ιταλία. Και αυτό θα πρέπει να έχει άποψη για το τι πρέπει να γίνεται στον άξονα Ανατολή Δύση και Βορρά Νότου. Μιλήστε μαζί του και πείτε του και εσεί δύο λόγια. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ελπίζω, προσωπικά το λέω αυτό, ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούν να κάνουν κάτι. Όχι όμως να υπάρξει ένα ειδικό ταμείο, να κοιτάζουν το θέμα της διασύνδεσης διασυνοριακά ευρύτερα. Και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής θα με πυροβολούσε αν έλεγα να γίνει ένα ειδικό ταμείο. Έχουμε ρόλο διασυνοριακά, έχουμε ρόλο ε, συντονιστικό, αλλά δεν έχουμε λόγο στη χρηματο... δεν, δεν, έχουμε, δεν πρέπει να χρηματοδοτήσουμε. Χρηματοδοτούμε ένα κομμάτι του Τωρίνο Νοβάρα, αλλά μόνο εάν έχει κάποια ε, συμπληρωματικότητα η δική μα συνεισφορά. Ξέρω εγώ μια μελέτη σκοπιμότητα. Η Ιταλία είναι πλούσια χώρα. Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούμε εμεί το σύνολο. Κύριε Τικάου. Κύριε Τικάου. Κύριε Τικάου. Από εκεί πέρα είστε, αν κατάλαβα καλά, ε. Και θέλετε να συνδεθεί το 6 και το 17. Να σας πω την αλήθεια, εμένα το 6 με ενδιαφέρει. Το σημείωσα ωστόσο. Θα δω και με τους συναδέλφους του 17, αν έχετε κάποια καλή πρόταση να μας το πείτε. Ευρώπη είναι και το Βουκουρέστι, κάπως πρέπει να συνδεθεί. Ας πείτε λίγο τα μαλλιά μου. Τέλο πάντων, θα ζήσω μερικά χρόνια ακόμα. Να φτάσουμε στη Βουδαπέστη και βλέπουμε. Τι... Σας είπα ότι δεν έχουμε σταματήσει τίποτα, υπάρχουν ωστόσο οι περιφερειακές εκλογές και περι... Ε, περιμένουμε το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να με βοηθήσετε απευθυνόμενοι στην τελική κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει το κομμάτι της ε, κοιλάδας της Σούσα ε, μετά τις εκλογές. Όντως κύριε Βανμπάλε, το κράτος είναι κυρίαρχο. Άρα ο κίνδυνος εδώ είναι η επανεθνικοποίηση οτιδήποτε. Τραπεζών, υποδομών κλπ. Θα συμφωνήσουμε φαντάζομαι εδώ. Τώρα, κόπερ τη βάτσα. Τι γίνεται, γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Κάποτε υπήρχε ένα άνθρωπο που τον έλεγαν Τίτο. Ο Τίτο πριν από πολλά χρόνια κατέλαβε την Τεργέστη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και είναι ακόμα ένα θέμα μεταξύ Ιταλίας και Ιουγκοσλαβίας. Το κόπερ είναι ένα μεγάλο κομμάτι, πολύ σημαντικό γιατί είναι το μόνο λιμάνι της Σλοβενίας. Δίπλα στην Τεργέστη. Εμείς θέλουμε να υπάρξει σύνδεση της Ντιβάτσα και με την Τεργέστη και με το Κόπερ και να γίνει αυτό με τρόπο θετικό και για τις δύο χώρες. Όπω ξέρετε εγώ δεν εμπλέκομαι, δεν, έχω, δεν παίρνω θέση. Και οι δύο περιοχέ είναι πανέμορφες. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι η ιστορία δεν μπορεί να καθορίζει το μέλλον. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια κοινή δομή και η κοινή δομή θα είναι στην Τεργέστη. Με Σλοβαίνου και Ιταλούς. Ο Υπουργό Μεταφορών τη Σλοβενία είναι ένα νέο. Τα μισά μου χρόνια έχει. Υποσχέθηκε να το κάνει. Πιστεύω ότι μια τέτοια νέα προσέγγιση χρειαζόμαστε. Εξαετή απόσταση είναι 600 μέτρα. Ε, μάλλον, ε, συγγνώμη, το, η υψομετρική διαφορά είναι 600 μέτρα. Η Τεριές είναι στη θάλασσα, η Λιβάτσα είναι στα 600 και ακόμα πιο πάνω είναι η Λουμπλιάνα. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια ε, μορφή σύνδεσης που να είναι εφικτή γερμανικά. Τώρα, για τον κύριο Ντοτά. Πρέπει να καταλαβαίνω την γαλλική άποψη. Χαίρο για την κυβέρνηση, της, για την υποστήριξη της κυβέρνησης, αλλά δείτε και τα προβλήματα που έχουν αλλού. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε αγαπητέ κύριε Μπριγχόρστ... Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Άμα λες λέει το πρόβλημά σου, το ξεφορτώνεσαι κατά το ίμιση. Έχουμε βέβαια και τον υπτάμενο Σκοτσέζο το πρόβλημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Και έξω ονόματος της Επιτροπής. Προσβλέπουμε και στη μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. If we can now uh, move on to the να προχωρήσουμε. Στο 1 και 17. Mr. Reuter is it who's coming up to do those. This is the Berlin Milan. Μιλάμε για την γραμμή 1. Βερολίνο, Μιλάνο, Παλέρμο. Ο κ. Βαν Μίρτ ήταν ο συντονιστή, τον ξέρουμε, ο οποίο δυστυχώ δυστυχώς και τραγικά χάθηκε πέρσι το καλοκαίρι, μεγάλη απώλεια. Τον θυμόμαστε. Το, η άλλη γραμμή που μας ενδιαφέρει εμάς τους βουλευτές πάρα πολύ είναι Παρίσι, Στρασβούργο, μια μικρή πόλη κάπου στην Αυστρία που τη λένε Βιέννα, μέχρι την Πρατισλάβα. Ο κύριος Ρόιτερ, 10 λεπτά. 10 λεπτά, δύο διάδρομοι, πρόεδρε. 5 λεπτά ο διάδρομος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, είναι λυπηρός ο λόγος που με φέρνει σε αυτήν εδώ την ε, θέση. Ο Κάλβαν Μίρτ ήταν ο συντονιστής ε, για το project Προτεραιότητα 1 από το 2005 και μετά. Εγώ ως ε, διευθυντής υπεύθυνος για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 1998-2000 ήμουν μέρος της Τριμερούς Επιτροπής που ασχολείται με το τούνελ Μπερναμπές πριν από μερικά χρόνια. Ο προκάτοχός μου επίσης ε, παρακολουθούσε αυτό το project για 20 χρόνια περίπου. Είναι λοιπόν λύπη από τη μία αλλά και χαρά που με κάνει ε, σήμερα να σας παρουσιάζω εδώ το πνεύμα αυτής της έκθεσης. Το βασικό μήνυμα είναι ότι το ένα προχωρά καλά και στα τρία κράτη-μέλη, Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία. Στη Γερμανία τα βασικά τμήματα που έχουν οριστικοποιηθεί αφορούν ε, το Βερολίνο Χάλε Λιψία και το άλλο είναι στο Μόναχο. Υπάρχει η συμφόρηση το σημείο ε, λειψία. Ε, έχουμε επενδύσει 7 δις που έχουν κινητοποιηθεί στην Ιρεμβέργη, στην Αυστρία και πάλι υπάρχει η κοιλάδα του ΙΝ που είναι ε, μια επένδυση 2,3 δις και το κομμάτι μεταξύ το Virgil και Innsbruck που αν κατάλαβα καλά στο τέλος του 2012 θα ανοίξει. Είχαμε την εναρκτήρια τερετή στην Ιταλία μεταξύ Βερόνα Μπολόνια και Μιλάνο Μπολόνια που είναι και κινητήριες δυνάμεις για αυτό το project. Και θα γίνουν και τα εγγένεια Μπολόνια ε, Φλωρεντία μέχρι το τέλος του 2009. Η Ιταλία λοιπόν εκτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του ένα και δημιουργεί τη ραχοκοκαλιά του δικτύου υψής της ταχύτητας στην ε, Ιταλία. Αυτά είναι τα καλά νέα. Ο Καρλ Βανιέτ ε, όμως ξεκάθαρα επικεντρωνόταν σε αυτά τα θέματα που ήταν τα πιο δύσκολα. Και από την αρχή ο συντονιστής είχε ταυτοποιήσει ε, το σημείο διπλής ε, διασυνοριακής ε, προσπέλασης μεταξύ Μονάχου και Βερόνας ήταν ένα προβληματικό θέμα. Εκεί υπάρχουν βασικά θέματα, η Σύρακα Μπερναμπές και ο Βόρειος και Νότιος Άξονας. Εδώ βέβαια ένα καλό νέο είναι ότι η αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει ολοκληρωθεί για το τούνελ και Περιμένω τις ερωτήσεις της κυρίας Λίχτενμπέργκερ γι' αυτό. Και ε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Από την Αυστριακή και Ιταλική πλευρά, τον Ιούλιο του 2009 είχαμε και οικονομική και τεχνική έγκριση για το τούνελ. Η κατασκευή λοιπόν της σύραγγας ε, πρέπει λογικά να ξεκινήσει το 2010 και να τελειώσει μέχρι το 2022 που είναι πολύ αργότερα από ό,τι θεωρούσαμε αρχικά όλοι. Ταυτόχρονα όμως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξεκινά αυτή η δουλειά. Την ίδια στιγμή, και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, Αυτές ε, οι συνδέσεις, η, ε, η όπως λέγονται στα γερμανικά, είναι οι, οι περιοχές όπου χρειαζόμαστε οικονομικές εγγυησει επίσης ε, να χρησιμοποιείται η νέα γραμμή Granarel σε όλη τη δυναμικότητα να υπάρχει διαλειτουργικότητα της υποδομής και αυτό δεν είναι μόνο το ERTMS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης των Συντηρονομικής Κυκλοφορίας, αλλά αυτό να ισχύει και για το μήκος των ε, αμαξοστοιχειών ε, και τα βάρη και των συστημάτων και τα συστήματα γενικότερα. Επίσης, να σας πω με χαρά μου ότι ο Καρλ Βίνκε που εργαζόταν στο ERTMS έγραψε μία επιστολή πρόθεσης ε, για τον διάδρομο Β του ERTMS ε, που είναι ταυτόσιμος ε, με το project προτεραιότητας που συζητάμε. Τέλος, ο Καλ Βαν ήταν ιδιαίτερα δραστήριος ως προς το να διασφαλίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία γιατί ε, το, η πλατφόρμα εργασίας και η ομάδα εργασίας Brenner έπρεπε να φτιάξουν ένα σχέδιο δράσης που θα είναι και αυτό διαθέσιμο. Υπάρχει μια κοινή δήλωση που υπογράφηκε στη Ρώμη από τους παλιούς ενδιαφερόμενους με την εξαίρεση ενός, ίσως θα σας πω κάποια πράγματα γι' αυτό αν χρειάζεται ήταν, το, ήταν γερμανική σιδηρόδρομη Deutsche Bahn εξαιτίας της αλλαγής ε, της ανώτατη διοίκηση που έλαβε χώρα εκείνη την εποχή. Αυτό το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 50 επιμέρους μέτρα που θα πρέπει να συμβάλλουν στην έγκαιρη εκτέλεση του βασική της βασικής σύραγγας εσείς στο Κοινοβούλιο συμφωνήσατε να υπάρξει νέο συντονιστή ε, για το Project 1. Το όνομα παραμένει βέβαια ανοιχτό, πρέπει να ελεγχθεί και εξαιτία των γερμανικών εκλογών δεν έγινε ως τώρα. Όμως ε, είμαι πεπισμένος ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα εργαζόμαστε όλοι υπό το πνεύμα του Καρλ Βαν Μίερς ε, ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το project. Αυτά για το 1. Να περάσω στο 17 αμέσως. Αυτό το έργο, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα έργο όπου είχαμε τον Πίτερ Μπάλας ως συντονιστή. για έναν πολύ καλύτερο λόγο δεν βρίσκεται εδώ. Είναι υπουργός εξωτερικών της Ουγγαρίας αυτή τη στιγμή. Έχει και όμως μια, και μια τεχνική διάσταση η θέση του. Ελπίζουμε ότι θα επανέλθει βέβαια σε αποκλειστικά ευρωπαϊκά θέματα, όχι μόνο στα ευρύτερα διεθνή θέματα. Το έργο από μόνο του είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Από τη γαλλική πλευρά έχουμε το κομμάτι της σύνδεσης, όχι ακριβώς στο Στρασβούργο ακόμα, πηγαίνει στον Ποντλεκούρ. Είμαστε όμως στη δεύτερη φάση. Η γέφυρα του Κέλ μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας είναι υποκατασκευή. Ε, διευκολύνει όχι μόνο τις, σιδηροδρομική, ε, τις μεταφορές αλλά και τις μεταφορές ε, στο Ρήνο. έχουμε λοιπόν καλύτερη πολιτική για, τους, υδάτινους, για τις υδάτινες οδούς. Όφενμπουργκ Καλσρούι επίσης, Καλσρούι Στουτκάρδη, Στουτκάρδη Ούλμα θα ξεκινήσει μεταξύ του 2010-2020 και η οριστικοποίηση του τμήματος Augsburg Μόναχου θα γίνει το, μέχρι το τέλος του 2010. Θα γίνουν συζητήσεις στη Γερμανία τους επόμενους μήνες ε, σχετικά με την εκτέλεση του τμήματος αυτού μεταξύ Ούλμ και Augsburg. Ε, Θεωρούμε όμως παρόλα αυτά ότι προχωρεί ικανοποιητικά το ζήτημα. Η Αυστρία φτιάχνει πολύ γρήγορα δύο σιδηροτροχές από το Λίντ στη Βιέννη που θα πρέπει να ξεκινήσει μέχρι το 2013 και θα κερδίζει κανείς 30 λεπτά μέχρι τη Βιέννη και 40 λεπτά από την Βιέννη στην Κροατία, στο τούνελ του Λάινσνεν, εκεί που θα δημιουργηθεί ένας νέος σταθμός μεταξύ του, ανατολ... του δυτικού σταθμού και του βασικού, του κεντρικού σταθμού. Στη Σλοβακία χρειαζόμαστε μόνο μερικά χιλιόμετρα για να συνδέσουμε τη Βιέννη με την Σλάβα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, θα γίνει η χρηματοδότηση της σωστής σύνδεσης και περιμένω με ανυπομονησία τις ερωτήσεις γι' αυτό. Αλλά για μένα, για να, είμαι, ε, να εκφράσω και την προσωπική μου γνώμη αν μπορώ να την πω, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σύνδεση που να περιλαμβάνει και τα αεροδρόμια. Να είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Λόγω της ε, πολιτικής διαλειτουργικότητας φυσικά. Ο Πίτερ Μπάλλας ε, ε, κατά τη διάρκεια της θητείας του έκανε τα πάντα για να μπορέσει να έχει επιστολή πρόθεσης και από τα τέσσερα κράτη-μέλη. Έχουμε τη δήλωση υποστήριξης από πάνω από 100 οικονομικές και δαφικές οντότητες. Υπάρχουν επίσης διασυνοριακές συμφωνίες μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το project ε, μπορεί να θεωρείται κάτι σαν παραδειγματικό έργο, δύσκολο, με πολλές δυσκολίες. Όπως έλεγε ο κύριος Μπριγχορτς και πριν, το κάθε έργο είναι πολύ καλό όταν το κοιτάς γενικά, όμως τελικά υπάρχουν επιμέρους προβλήματα που ε, αναδύονται και εκεί οι συντονιστές παίζουν σημαντικό ρόλο, διασφαλίζουν ότι προχωρούν τα project. Αυτά μπορώ να σας αναφέρω. Δεν είμαι συντονιστής, ούτε έκανα αίτηση για αυτή τη θέση. Βρίσκομαι εδώ δυστυχώς ε, ε, λόγω της απώλειας του Καλ Βαντερμίν και ε, ως αντικαταστάτης του Πίτερ Βάλλας. Θα χαρώ να δεχθώ τις ερωτήσεις και του συναδέλφου Χέραλ, και ο συνάδελφος Χέραλτ Ρόιτερς επίσης θα μπορέσει και αυτός ενδεχομένως να απαντήσει τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε κυρία Γέγκερτ προς το παρόν έχει ζητήσει το λόγο, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλοι. Θα τις ε, κάνουμε όλες μαζί ε, για όλα τα project και μετά μπορούμε να χωρίσουμε τις απαντήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Κιν για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι άξονες έχουν ε, ως ε, στόχο να μεταφέρουν τις περιοχές ε, στόχους την κυκλοφορία. Αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη, ε, βόρεια και νότια και αριστερά και ανατολή-δύση έχουν προβλήματα με τη σύνδεση. Ας πούμε το τούνελ Μπρένερ ε, εκτελείται ε, σε μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλές, πολλά συνοριακά προβλήματα και είναι σημαντικό να έχουμε από τη Βρένη στην ε, Αυστρία και στο Μόναχο και ε, προς τα κάτω Βρένη ε, Βερόνη, Βερόνα να έχουμε καλή διανομή της κυκλοφορίας γιατί η κυκλοφορία εκεί συνδέεται άμεσα με τους δρόμους που πηγαίνουν βορρά-νότο. Έτσι λοιπόν έχουμε δρόμους ε, που ε, διασχίζουν όλη την Ευρώπη και δεν σταματούν κάπου. Όταν ε, πάει κανείς από το Παρλέμρμο στο Βερολίνο βλέπει πώς δικτυώνονται οι διασυνδέσεις. Έχουμε σύνδεση με το 6, διευρωπαϊκά δίκτυα νούμερο 6. Εκεί είχαμε προβλήματα με την διάσχιση των Άλπαιων Και εδώ είναι το ερώτημα πώς γίνεται η δικτύωση, η διαδικτύωση. Ε, πώς ε, περνάει κανείς από τις ε, Άλπεις και θέλει να πάει προς την Αδιαρατική, από τον Κράτς και θέλει να φτάσει στη Βαρσοβία ή στην Πράγα και στο Βερολίνο. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξεκινάμε από το Βερολίνο και να πηγαίνουμε προς την ε, Αδριατική και γενικά ε, προς την Ανατολή και τη Δύση. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι άξονες να, να μην είναι μικροί, αλλά να φτάνουν μέχρι και τη Σκανδιναβία αν είναι δυνατόν. Κυρία Μάισερ, ευχαριστώ καταρχάς για την παρουσίασή σας. Έχω δύο ερωτήσεις, είμαι καινούρια, ίσως οι παλιοί να τα ξέρουν, αλλά για το βασικό τούνελ ε, Βρένης ε, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ε, για, την, για το πόσο έχει σχεδιαστεί σωστά και πόσο αναγκαίο είναι, είναι η ερώτησή μου. Επίσης, όταν περάσει η κρίση θα αυξηθεί η μεταφορά όμως δεν είναι αρκετό τελικά το ε, τούνελ αυτό, ε, όπως λένε. Μετά, κάτι που δεν κατάλαβα. Είπατε ότι στη σύνδεση Βιέννη-Βρατισλάβα, που είναι μικρή απόσταση, χρειάζεται κάποιος μερικά χιλιόμετρα μόνο. Ε, και δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε τη σωστή γραμμή, είπατε. Όμως τι είπατε τελικά εσείς, πρέπει να μπουν και τα αεροδρόμια μέσα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Βιέννη, Μπρατισλάβα και μαζί και τα αεροδρόμια ή τι άλλο. Ποια είναι η εναλλακτική για τη χάραξη αυτής της γραμμής. Επόμενος. Βαθιά Ευχαριστώ πολύ. Εξαιτία του χρόνου θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο βέβαια. Το βασικό, η βασική σειρά βρένει. Έχουμε πει ότι υπήρχαν ε, κάποιες κάποια εξέταση για το πόσο αντέχει αυτό. Υπήρχαν γεωλογικά προβλήματα στη νότια πλευρά. Όσα έγιναν στο παρελθόν σχετικά με το γεωλογικό ρίσκο, ε, στο παρελθόν όσα υπόθηκαν έχουν περάσει υπάρχουν ΣΔΙΤ ε, ε, στην ε, Ιταλία και στην Αυστρία και υπάρχει και εμπλοκή του κοινού εκεί. Υπάρχει και θέμα των πόρων σε κάποιες περιοχές εκεί. Σε αυτό το project έχω τη δυσκολία ότι σύμφωνα με την έκθεσή σας ε, για την νότια σύνδεση μέχρι τη Βερόνα υπάρχουν και άλλα projects και με εκπλήσει που οι Γερμανοί στο σχέδιό τους δεν έχουν βάλει ως προτεραιότητα την ε, διοχέτευση προς ε, το τούνελ Μπρένερ. Αυτό είναι η βασική, το βασικό θέμα. Οι μεταφορές που έρχονται από τον ε, Νότο ή τον Βορρά δεν θέλουν να πάνε στο Ινσπουργκ, θέλουν να πάνε από τις Άλπεις. Όταν αυτό το κομμάτι μεταξύ Μπρένερ και Βερόνα ε, έχει τέτοια καθυστέρηση και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, πολύ πολύ πλοκές διαδικασίες ε, κατασκευής ε, δεν μπορούμε να συζητάμε για το τούνελ και για τις εγγυήσει ε, Ιταλίας θα ήθελα να το συζητήσουμε ξεχωριστά γιατί ως τώρα δεν είναι αξιόπιστο αυτό που έχουμε. Τελευταίο σημείο, μιλήσατε για τη διαλειτουργικότητα από τεχνική πλευρά. Εγώ πάω ένα βήμα παραπέρα. Ξέρω ότι πολλά τρένα παραμένουν στο Βρένερ γιατί θέλει να δει για την Ιταλία και αυτό ε, είναι δύσκολο γιατί χρειάζονται δύο μηχανές για να συνεχίσουν και είναι για μένα σημαντικό γιατί εκεί έχω μεγαλώσει. Τώρα για τη Μεσίνα. Έχει ενημερωθεί αυτό το κομμάτι του project από την Ιταλία, η γέφυρα δηλαδή εκεί δεν ξέρουμε ακριβώ πώς έχει η κατάσταση. Για το διάδρομο 17, ποιο από τα τρία project είναι ε, δυνατό. Υπάρχουν τρει εναλλακτικέ, δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Εγώ θα ήθελα να, ε, κάτι που να γίνει γρήγορα και μετά να πάμε από πάνω ε, το από πάνω κομμάτι που θα μπορέσει να γίνει ακόμα πιο γρήγορα. Για τον 17 επίσης ο κύριο Μπάλας είχε πει ότι υπάρχουν εναλλακτικέ μεταξύ Μονάχου και Λίντς ε, γιατί υπάρχει εκεί και το βιομηχανικό τρίγωνο, το χημικό τρίγωνο και μπορούμε να το ε, συνδέσουμε και αυτό και θα ήταν έξυπνο να γίνει γιατί υπάρχει και μεταφορά εμπορευμάτων από εκεί. Και τέλος, τι γίνεται με τη Γαλλία, έχουμε και μεταφορά εμπορευμάτων ή έχουμε απλώς ε, τα ΤΖΒ για τα ε, μεταφορά επιβατών. Για τα εμπορεύματα λοιπόν υπάρχει κάτι που έχετε σκεφτεί ε, για τη χρήση των παλιών γραμμών. Ευχαριστώ. Άλλοι τέσσερι έχουν ζητήσει το λόγο. Κόνιτσεκ πρώτος. Ο κύριο Κόλιτσεκ πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ επιγραμματικός. Μου αρέσει να μιλάω για όλους αυτούς τους διαδρόμους και τις διάφορες διαδρομές. Η τσεχική δημοκρατία όμως είναι μια μαύρη τρύπα. Τίποτα δεν διασχίζει τη χώρα. Ο πρώτος ομιλητής είπε ότι πρέπει να διασχίσεις και την Τσεχία σε κάποια φάση. Και αν θέλω να περάσω και να πάω βόρεια της Βιέννης, πάλι πρέπει να περάσω κάποια χώρα. Μιλάμε για τον Περνό, τον Περνό που είναι στην ε, Τσεχική Δημοκρατία και την Πράγα που είναι στην Τσεχική Δημοκρατία. Αυτοί που ασχολούνται με τους σιδεροδρόμους ίσως θεωρούν ότι το μόνο που πρέπει να κάνουμε δεν θα, είναι, θα, θα ευρεί άλλη λύση και όχι μέσω των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων. Ρωτάω, θα υπάρξουν οι αναγκαίες διασυνδέσεις. Πάντα συνδέουμε το α με το β. Μέχρι τώρα όμως δεν μπορέσαμε να κατασκευάσουμε τα 880 μέτρα που θα συνέδεαν τη νέα γραμμή με τις παλιές. Τι θα συμβεί λοιπόν, αυτά που ανέφερα, Πρέτσλαβ, Βιέτσιν, υπάρχει ένας διάδρομος που κατασκευάζεται αλλά στο Γέτσιν υπάρχει μία σύραγγα με μία μονογραμμή. Και πίσω τον Τιέτσιν, στην κοιλάδα, ξανά μόνο μία γραμμή έχουμε που πάει στη Δρέσδη. Δηλαδή όλα είναι πολύ στριμωγμένα και στενά αυτή την Μορα... τη Μοραβία δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διασύνδεση προς Πολωνία βόρεια του Μπρέτσλα υπάρχει διάδρομος αλλά μέχρι 160 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για ράγες χαμηλότερης ταχύτητας, όχι για τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Κυρία Γέγκλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δεν είμαι μέλος εδώ και 10 χρόνια και μπορώ σήμερα να μιλήσω για τον διάδρομο 17. Αντίθετα με την ερώτηση και ο κύριος Κράμερ θα μιλήσει μετά, στη δίκαιη επικριτική ερώτηση για διάφορα θέματα όπως πώς θα συνεχίσουμε. Σήμερα βρίσκομαι εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάλας. Ο κύριος Μπάλας έχει κάνει γι' αυτό το κομμάτι της Γερμανίας για το οποίο μιλάμε πετύχει το κατόρθωτο. 15 χρόνια στη Γερμανία συζητήσαμε για το πώς θα γίνει χρηματοδότηση ε, για τη Στουτκάρδη και γενικά της Άλπης. 15 χρόνια μέσα στη Γερμανία υπήρχε αυτή η συζήτηση. Το άντεξε αυτό όμως στις 2 ε, Απριλίου 2009 η Περιφερειακή και Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και από την Deutsche Bahn έχουν υπογράψει. Αυτό ήταν μεγάλο επίτευγμα. Αυτή τη στιγμή βέβαια παραμένουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Και από, έρχομαι, από εκεί που προέρχομαι εγώ, από το Όμπερ υπήρχε κριτική ότι ε, γιατί πληρώνουμε για πράγματα που δεν μας αφορούν. Σήμερα στο νότιο κομμάτι μέχρι την κοιλάδα του Χίντεφτερ υπάρχει ε, αυτή η αναγνώριση ότι αυτή, αυτός ο διάδρομος είναι ραχοκοκαλιά. Μέσα λοιπόν από αυτή την ε, συνολική άποψη βρίσκομαι εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάλας ε, και παρακαλώ αυτούς που θα έρθουν στο μέλλον να γνωρίζουν ότι χρειαζόμαστε αυτή τη γραμμή και ε, αν στο τέλος θα γίνει Παρίσι, Βουδαπέστη και αν θα υπάρχει ε, δια και χρήση πολλών μέσων, αυτό το προσυπογράφουμε Κύριε Κράμερ, τώρα έχετε κι εσείς ε, ε, για τη Στουτκάρδη παλέψει στις ε, εκλογές ως πράσινος. Εγώ τουλάχιστον εδώ είμαι εδώ για να μιλήσω για επιτυχία. Ελπίζω να συνεργαστούμε ώστε να έχουμε και άλλες επιτυχίες. Ευχαριστούμε, Μίχαλ, έχεις το λόγο. Αν θέλεις να το κάνεις μέσω του Προέδρου, βέβαια δεν έχουμε πρόβλημα. Να ξεκινήσω με το Βερολίνο Στοκχόλμη. Έχω εδώ στα έγγραφά μου έναν ε, διάδρομο ο οποίος πρέπει να πάει προς τα πάνω. Βερολίνο, Κοπενχάγη, Στοκχόλμη. Όμως ε, υπάρχει και το Βερολίνο, Αμβούργο, Κοπενχάγη. Εχθές ζητήσαμε για τους εννέα διαδρόμους για τη μεταφορά ε, εμπορευμάτων η οποία δεν θα περάσει από το Βερολίνο, από Ίνσπουργκ, Αμβούργο, Κοπενχάγη, Στοκχόλμη. Στα διευρωπαϊκά δίκτυα λοιπόν έχουμε τρεις διαφορετικές επιλογές. Τι ισχύει τελικά. Θα ήθελα τελικά να βρείτε μία ε, ενιαία θέση, να μην έχουμε αλλού στα ένα χαρτί το ένα και σε άλλο χαρτί το άλλο, γιατί δεν θα έχουμε καθόλου χρήματα στο τέλος για τίποτα. Τώρα για το αγαπημένο σας αυτό project, κυρία Γέκλερ, υπήρχαν κάποιοι συντηρητικοί από τη Βάδη Βιτεμβέργη με τους οποίους ε, συμφωνούσα. Έλεγαν ότι όλα τα λεφτά πάνε στη Στουτκάρδη. Στην, ε, οι πράσινοι ήμασταν ισχυροί στη Στουτκάρδη εξαιτία των θέσεών μα. Δεν θέλουμε να δίνουμε ούτε ένα σεντ στην Ευρώπη. Ε, από την Ευρώπη να έχουμε ίδια χρηματοδότηση. Όλα τα χρήματα που δόθηκαν για τη Στουτγκάρδη βασίζονται σε δεδομένα του 2004. Από το 1998 συγκεκριμένα προέρχονται αυτά. Ε, αυτό είναι γερμανικό θέμα. Γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσε ποσοστιαία χρηματοδότηση, αλλά συγκεκριμένα ε, κόστη. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, όταν έχουμε τη διαδρομή στις Άλπεις και πάλι ε, θα έχουμε από το Σουτκάρδι 21 στις Άλπεις ε, και πάλι δεν θα έχουμε πολλά ε, εμπορεύματα που θα περνάνε εκεί. Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη η δυναμικότητα αλλιώς γιατί δίνουμε τόσα λεφτά. Πραγματικά εδώ με ρέθησε η κυρία Γέγκλερ. Ε, για τη Βιέννη ένα πράγμα θα πω. Με τον κύριο Μπάλα συζητήσαμε πολύ συχνά ότι οι Σλοβάκοι θέλανε τρία πράγματα, τελικά πήρανε ένα, το αεροδρόμιο. Άκουσα επίσης ότι δεν θα γίνει άμεση σύνδεση ε, μέσα από τη Βιέννη ε, κατευθείαν στο αεροδρόμιο, αλλά πρέπει κανείς να αλλάξει. Αυτό θα ήταν τρελό. Και αυτό θα ήταν εθνικό θέμα, όχι διευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, τι χρησιμοποιεί λοιπόν ένας νέος σταθμός ο οποίος έχει χρηματοδότηση 3% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά μπορεί να μην είναι λειτουργικός γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που το χρησιμοποιεί και τελικά ε, είναι μη λειτουργικός. Λοιπόν, ε, πείτε μας τελικά τι γίνεται στη Βιέννη. Μπορείτε είχατε πει από την αρχή αυτά. δεν θα ξοδεύαμε 15 λεπτά. Η κυρία Ράνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι πιο σύστημη. Αλλά δεν θα αφήσω την ευκαιρία, αφού σήμερα μιλάω για πρώτη φορά ως διάδοχος του Reinhard Rank στον διάδρομο αυτό. Να συμφωνήσω με τον κύριο Κούν είναι σημαντικό αυτός ο βαλτικός αδριατικός διάδρομος να μην έχει μόνο σύνδεση ε, βορρά-νότου αλλά και ανατολής-δύσης. Με αυτόν τον διάδρομο μπορούμε να ε, διευκολύνουμε άλλες συνδέσεις ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μέσω της σύνδεσης των σιδηροδρόμων. Αυτό είναι ίσως ε, το πιο ακριβό project. Ε, έχει ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί το 2015. Ε, δεν ξέρω κυρία Λιχτενμπέργκερ τι είπατε, δεν το θέλετε. Εκτός μικροφώνου κυρία Λιχτενμπέργκερ. Um Εδώ δεν είναι δική μας δουλειά να βρούμε τα λεφτά. Κυρία Λιχτεμπέργκερ, δεν έχω πρόβλημα να απαντήσετε, αλλά να απαντήσετε μέσω του Προεδρείου για να ξέρουμε τι λέτε. Σύντομα, να πω ότι υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον για αυτόν τον διάδρομο, γιατί πραγματικά φαίνεται ότι είναι σημαντικός. Ο βασικός σταθμό, ο κεντρικό σταθμό στη Βιέννη σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερη σημασία. Ε, project που χρειάζεται προτεραιότητα και ελπίζω να ε, ακούσετε και σήμερα και τις πληροφορίες που έχουν να δοθούν για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχω ένα απλό ερώτημα. Κύριε Ρότλε, περίπου 25 δισεκατομμυριάκια θα κοστίσει. Αν μπορεί να φτάσει ο διάδρομος μέχρι το Μάντσεστερ, είναι κάτι προσωπικό, ένα ερωτηματάκι έχω. Ευχαριστώ. Πάντα πρέπει να απαντά κανείς πρώτα τα ερωτήματα του Προεδρού. Αν μας να βρούμε τα χρήματα, ναι, μπα καταφέρουμε. Το να περάσουμε το Παρίσι είναι το πρόβλημα, συνεχίζει χαριτολογώντα ο Πρόεδρος. Πολύ γρήγορα να προσπαθήσω να απαντήσω στι ερωτήσεις. Πολλέ από τι ερωτήσεις δεν θα βρούνε σίγουρη απάντηση, αλλά θα τις διαβιβάσω στους μελλοντικούς συντονιστές τα ερωτήματα. Κύριε Κούν. Για να απαντήσω στη δική σας ερώτηση και αυτό είναι μια ερώτηση που ε, έχουμε συζητήσει και με την κυρία Ράινερ. Πρέπει η μελλοντική συζήτηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα να μπει στο πλαίσιο για ε, τη συζήτηση για επιπλέον διαδρόμους και να δούμε πώς θα τεθούν οι προτεραιότητες ε, μεμονωμένα ώστε να φτιάξουμε ένα συνεκτικό δίκτυο το οποίο ε, θα, έχει, ε, θα συνάδει με την πολιτική μεταφοράς. Και αυτό έχει να κάνει με το συνολικό ερώτημα της διαδικτύωσης με την Βόρεια Θάλασσα, με την Σκανδιναβική περιοχή και με τη Μεσόγειο μέσα από το βασικό τούνελ του Μπρένερ. Κατά τα άλλα να πω ξεκάθαρα, κυρία Μάισνερ, ότι σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις ε, και στην παλιά και στην καινούρια, ε, και στο καινούριο κομμάτι ε, έχουμε περίπου 400 οχήματα την ημέρα, μεγάλο ποσοστό λοιπόν μεταφοράς μέσων μεταφοράς και αυτό είναι πραγματικά πρόκληση για αυτό το project. Κύριε Κούριτσεκ, μιλήσατε για την κατάσταση στην Τσεχία, στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Φαίνεται, ε, το είπε και η κυρία Τικάου πριν, Μάλλον ο κύριος Κράμερ έκανε την ερώτηση επίσης πώς καταφέρνουμε τη διασύνδεση με την ε, ε, Ανατολική Ευρώπη. Μιλήσατε για το 17 ε, και είπατε ότι το πρόθεσε ως εκεί ο κύριος Μπάλαστ. Να πω προς υπεράσπιση του ότι υπάρχει το 22, project 22, το οποίο ακριβώς φέρνει αυτή τη διασύνδεση και με την Τσεχία και, και με την Βουδαπέστη μέχρι το Βουκουρέστι. Και πριν γίνει υπουργό ε, Εξωτερικών, ο κύριος Μπάλας, μου είχε πει ότι πρέπει να είμαστε βέλικτοι με τους κανόνες έτσι ώστε να προωθήσουμε και το Project 22. Από αυτή λοιπόν την άποψη έχουμε την ίδια κατεύθυνση. Κυρία Λίχτεμπέργκερ, θέσατε πολλές ερωτήσεις. Σημειώνω ότι υπάρχουν ακόμα κάποια γεωλογικά προβλήματα τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε. Να πω βασικά ότι ο Ευρωπαίος Συντονιστής οι συντονιστές, οι Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε και το θέμα της επικουρικότητας, γιατί πολλά από αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο. Και πρέπει κατά κάποιο τρόπο να δούμε πού είναι απαραίτητη η Ευρώπη, πού είναι χρήσιμη η Ευρώπη και από την άλλη να δούμε ταυτόχρονα πώς λειτουργούν τα πράγματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και πώς προχωρούν. Συμφωνώ πλήρως και απολύτως ε, για το θέμα των ε, διαδρόμων διοχέτευσης. Δεν μπορείτε να έχετε τη σύραγγα και να μην έχετε τις οδού που οδηγούν εκεί, Αυτό είναι ο βασικός ρόλος των συντονιστών. Να διασφαλίσουν ότι ταυτόχρονα με την κατασκευή της σύραγγα υπάρχει και η κατασκευή των οδών που οδηγούν εκεί, είτε είναι στο Μόναχο είτε οπουδήποτε. Είτε είναι σύνδεση σε αεροδρόμιο, είτε στο τρίγωνο των χημικών βιομηχανιών, είτε υπάρχει διασύνδεση με την ε, Βερόνα και αν είναι σωστή εκεί η χρηματοδότηση. Τέλος πάντων αυτή είναι η δουλειά του συντονισμού. Αυτό είναι και στα πλαίσια του σχεδίου δράσης. Ε, αυτό που ορίστηκε ως αποστολή. Κυρία Μάισλερ, θέτωσατε το θέμα της Μπρατισλάβα. Για μας είναι ξεκάθαρο. Εμείς χρηματοδοτούμε μόνο το νότιο κομμάτι. Την νότια σύνδεση στο αεροδρόμιο. Αυτό είχε συστήσει ο κύριος Εμπάλας, αυτό εμείς χρηματοδοτούμε μέσα από τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα ήθελα για άλλη μία φορά βέβαια ίσως ε, να συζητηθεί το θέμα ώστε να έχουμε τη σωστή κατεύθυνση σε επίπεδο διαλειτουργικότητας. Κυρία Γέγκλε. Θα μεταβιβάσω στον κύριο Μπάλας αυτά που είπατε. Ήταν πολύ θετική η συμβολή. Και εμείς ε, ξεκάθαρα δεν μπήκαμε στο αντιφατικό θέμα του Στουτκάρδη, την οδό 21. Εμείς ε, προσπαθήσαμε να δούμε πώς εκεί θα λειτουργήσει η αρχή της επικορικότητας, το αν θα γίνει μέσω του 21 στη Στουτκάρδη είτε με κάποιον άλλον τρόπο, αυτό είναι κάτι που αφορά το κράτος ε, μέλος, δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Τώρα μέχρι την ερώτηση για το Μάντσεστερ νομίζω ότι έχω καλύψει. Ε, επειδή είναι ειδική ερώτηση χρειάζομαστε περισσότερο χρόνο γι' αυτό. Νομίζω κατά τα άλλα απάντησα στις ερωτήσεις σας. Α, για τη γέφυρα είπατε κάτι, ναι. Ναι, για τη γέφυρα. Είναι κομμάτι, ξεκάθαρα, και έτσι το ψηφίσατε στο Κοινοβούλιο, του Project 1. Είναι όμως επίσης ξεκάθαρο ότι δίνουμε προτεραιότητα στα διασυναριακά κομμάτια των διευρωπαϊκών δικτύων. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σίγουρα έχει σχέδιο για γραμμή υψηλής ταχύτητας από Μάντσεστερ για Λονδίνο. Ήταν κάπως αστεία αυτή η πρότασή μου, αλλά μπορεί να συμβεί τελικά. Απάντηση σε ερώτηση εκτό μικροφώνου. Ο Μάικλ είναι πολύ πιο εύκολο όταν είναι κανεί στην αντιπολίτευση. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι μια δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση εκ μέρου των δύο συντονιστών. Δυστυχώς έχουμε χάσει τον έναν. Ευχαριστώ τα μέλη. Τα ξαναλέμε στις 3 ακριβώς με τον κύριο Βαλέντε Ντιολιβέιρα θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα 21 για τους αυτοκινητόδρομους, τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους. Θα τα πούμε στις 3. Καλή σας όρεξη.